Λοιπόν, μπορούμε να υιοθετήσουμε την ημερήσια διάταξη αν κανείς δεν έχει αντίρρηση. Δεν βλέπω καμία αντίρρηση. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Ανακοινώσεις δεν υπάρχουν σήμερα. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία αφού προηγουμένως ελέγξουμε ότι υπάρχει απαρτία. Ελέγχουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Είμαστε εντάξει. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Έκθεση Μπάσεκουτ. Δόθεση της ενέργειας η οποία παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Ξεκινάμε λοιπόν. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Όπως θέλετε, μπορούμε να ελέγξουμε και ηλεκτρονικά. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Συν 19. Αγαπητοί συνάδελφοι, εγκρίνεται η συμβαστική 7. Ξέχασα όμως την κάρτα μου. Εγώ ψηφίζω όπως η ομάδα μου. Άλλη μία λοιπόν. Υπέρ ή κατά δηλαδή. Ακόμα και αν ψηφίσετε κατά. Η συμβαστική 7 περνάει. Περνάμε την προσθήκη στη συμβαστική 7 υπέρ. Τι συμβαίνει. Δεν ξέρετε τι να κάνετε. Τι συμβαίνει. Μην χαθείτε από τόσο νωρίς, γιατί είναι πολύ πολύ νωρίς. Είμαστε στην προσθήκη. Ευχαριστώ, Βίκτορα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Δεν εγκρίνεται με μία διαφορά, μία ψηφοδιαφορά. Και τώρα περνάμε στο άρθρο. Δεν δουλεύει εδώ το μηχάνημα. Δηλαδή ψήφισα, αλλά δεν ε, εμφανίστηκε. Κύριε Τέιλορ. Ήθελα να σας πω ότι ακόμα και αν ψηφίσετε υπέρ, είναι 18-18 και παρόλα αυτά δεν εγκρίνεται. Μπορούμε να ξαναψηφίσουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι 9 και 9 λεπτά. Μόλις αρχίσαμε. Υπάρχουν ε, κανόνες Θέλετε να ξαναψηφίσουμε. Μα το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Εντάξει. Ξαναψηφίζουμε προσθήκη στη συμβαστική 7. Δεν είναι δυνατόν να ψηφίζουμε και να ξαναψηφίζουμε στο ίδιο. Λοιπόν, τέλος της ψηφοφορίας. Τέλος. Υπάρχει ισοψηφία. Non. À mon avis, vous avez fermé le vote. Quand j'ai fermé le vote, j'ai... Τέλος της ψηφοφορίας. Τέλος. Τέλος της ψηφοφορίας, όποιος ήταν εδώ ψήφισε. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν με το άρθρο 102. Συγγνώμη, με την τροπολογία 102. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Το 102 απορρίπτεται. 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 6 περνάμε στην τροπολογία 110 υπέρ κατά αποχές η 110 απορρίπτεται. 2. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται η 2. 117 υπέρ. Κατά αποχές. Η 117 εγκρίνεται. Το πρωτότυπο κείμενο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται το πρωτότυπο κείμενο. Συνεχίζουμε με την 124 υπέρ. Κατά αποχές η 124 απορρίπτεται. 125 υπέρ. Κατά αποχές 125 απορρίπτεται. 119 και 128. Ψηφίζουμε από κοινού. Υπέρ. Συγγνώμη, την 119 και την 126. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. 19 υπέρ 19 κατά. Απορρίπτονται. Συνεχίζουμε. 127 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται η 127. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 129 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αλφα υπερ υπέρ αλφα κατά αποχές ψηφίζουμε ηλεκτρονικά 3α ψηφίζουμε Τέλος. Απορρίπτεται η 3α. 3β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Νομίζω εγκρίνεται παρόλα αυτά. Αρχή της ψηφοφορίας για την 3β. Τέλος. 20-19. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε. Συμβιβαστική 4. Κυρία Γιούτο. Συγγνώμη, δεν ε, λειτουργεί η κάρτα ψηφοφορίας μου. Να ψηφίσουμε σηκώνοντας το χέρι. Ψήφισα υπέρ στη συμβαστική. Άρα η 3β εγκρίνεται, λέει η Πρόεδρος. Μήπως μπορείτε να αλλάξετε θέση. Συμβαστική 4, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται η 4. Η 146, υπέρ, κατά, αποχές. 146 εγκρίνεται. 147 υπέρ. Κατά αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ελέγχουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται. Και συνεχίζουμε. Με τις ε, τροπολογίες που ακολουθούν μέχρι την 154, όλες μαζί υπέρ. Κατά αποχές ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτονται. Συνεχίζουμε με την 154. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η 154. 155. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται η 155 156 υπέρ κατά αποχές 156 γκρίνεται 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 160 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 161 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 162 υπέρ κατά αποχές 162 απορρίπτεται 163 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 164 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 165 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε Ψηφίζουμε την 165. Στους πράσινους κάποιος παραπάνω έχει ψηφίσει. Τώρα είναι εντάξει. Η 165 εγκρίνεται. 166. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 166. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Εντάξει. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Η 166 απορρίπτεται. Συνεχίζουμε. 192. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 195 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η 195. 198 υπέρ. Κατά αποχές αρχή της ψηφοφορίας επί της 198. Τέλος, η 198 απορρίπτεται. Η 28 υπέρ. Κατά αποχές Δεν είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. Αρχή της ψηφοφορίας ψηφίζουμε για την 28. Τέλος. Απορρίπτεται 28. 199 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 199 εγκρίνεται. Η 200 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 201 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 201 απορρίπτεται. 202. Α, να ελέγξουμε την 201. Αρχή της ψηφοφορίας για τη 201. Τέλος. Η 201 απορρίπτεται. 202 τώρα. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 203 κατά αποχές η 203 απορρίπτεται Α, να ελέγξουμε Αρχή της ψηφοφορίας Τέλος η 203 απορρίπτεται και περνάμε στη 208. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 208 απορρίπτεται. Α, ελέγχουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίζουμε για την 208. Τέλος. Η 208 απορρίπτεται. Η 209 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 209 απορρίπτεται. 210 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 210 εγκρίνεται. 211 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 211 απορρίπτεται. Η 33 υπέρ κατά αποχές θα επαληθεύσουμε αρχή της ψηφοφορίας για την 33. Τέλος. Η 33 εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε από κοινού την 34, 35 και 36. Υπέρ. Κατά αποχές. Οι τρεις αυτές τροπολογίες συγκρίνονται. Η 38 τώρα, υπέρ. Κατά αποχές. Η 38 απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Αρχή της ψηφοφορίας για την 38. Τέλος. Δεν εγκρίνεται. 20 ψήφοι κατά. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. να επαληθεύσουμε. Αρχή της ψηφοφορίας για τις 40. Τέλος. Η 40 απορρίπτεται. 41. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Η 41 απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά. Απόχες. Η 42 απορρίπτεται. Θέλετε να επαληθεύσουμε. Ας επαληθεύσουμε λοιπόν αρχή της ψηφοφορίας. 42 τροπολογία. Τέλος. Απορρίπτεται. Προχωράμε, προχωράμε. 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον απορρίπτεται. Αρχή της ψηφοφορίας. Επαληθεύουμε. Τέλος. Η 43 απορρίπτεται. 44 υπέρ. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, εγκρίνεται, συγγνώμη. 45 υπέρ κατά αποχές. Η 45 εγκρίνεται. 46 ψηφίζουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. Έτσι είναι πιο απλή η διαδικασία. Τέλος, η 46 εγκρίνεται. Συμβαίνουν και αυτά. 53. Ποιος είναι υπέρ της 53. Κατά. Αποχές. Η 53 εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Αρχή της ψηφοφορίας. 54. Τέλος. Εγκρίνεται 54. Συνεχίζουμε με την 56. Υπέρ κατά εποχές η 56 απορρίπτεται έχετε δικαίωμα θέλετε να επαληθεύσουμε αρχή της ψηφοφορίας τέλος η 56 απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα αρχή της ψηφοφορίας ψηφίζουμε την 57 τέλος η τροπολογία 57 εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται 58. 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται νομίζω. Θέλετε να επαληθεύσουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται η 59. Πρέπει να μου έχετε εμπιστοσύνη κυρία Γραπίνη. Και συνεχίζουμε με την 61 υπέρ. Κατά αποχές. Η 61 εγκρίνεται. Ναι, μπορώ να δεχθώ την ψηφοφορία αφού δεν τη ζητάει η κυρία Ρεποντάλων. Αρχή της ψηφοφορίας για την 61. Τέλος. Η 61 εγκρίνεται. Μα μπορείτε να μου έχετε εμπιστοσύνη. Συνεχίζουμε με την 62 υπέρ. Κατά. Απόχες. Η 62 απορρίπτεται. 63 υπέρ όχι συγγνώμη, 64 υπέρ κατά αποχές 64 εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές 65 εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 2 αρχή της ψηφοφορίας Τέλος. Η τροπολογία 2 απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά αποχές η 66 εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά αποχές η 69 εγκρίνεται. Α, θέλετε να ελέγξουμε. Η 70 υπέρ κατά αποχές. Η 70 Α, να επαληθεύσουμε. Αρχή της ψηφοφορία για την 70. Τέλος. Η 70 απορρίπτεται. 71. Υπέρ. Κατά αποχές η 71 εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές η 72 εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές η 73 εγκρίνεται Α, να επαληθεύσουμε αρχή της ψηφοφορίας Τέλος, η 73 εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 74 εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 75 Απορρίπτεται. 76. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 76 εγκρίνεται. 77. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 77 εγκρίνεται. 78. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 78 εγκρίνεται 79 υπέρ. Κατά αποχές. Η 79 εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στη 3 υπέρ. Κατά αποχές. Η 3 απορρίπτεται. Α, να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 3, αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος, η 3 απορρίπτεται. 81 υπέρ. Κατά αποχές η 81 εγκρίνεται. 80 υπέρ. Κατά αποχές η 80 απορρίπτεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 4 απορρίπτεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 83 εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 84 απορρίπτεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 85 εγκρίνεται. Η 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 86 απορρίπτεται. Α, να επαληθεύσουμε. Αρχή της ψηφοφορίας για την 86. Τέλος. Απορρίπτεται. Η 87 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 88 υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 88 εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 6 απορρίπτεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 89 εγκρίνεται. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται η 90. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 91 απορρίπτεται. 92 υπέρ κατά αποχές η 92 εγκρίνεται 93 υπέρ κατά αποχές η 93 εγκρίνεται 94 υπέρ κατά αποχές η 94 εγκρίνεται 95 υπέρ κατά αποχές Επαληθεύουμε. Αρχή της ψηφοφορίας ψηφίζουμε την 95. Τέλος. Εγκρίνεται η 95. Α, όχι, απορρίπτεται, λέει η πρόεδρος. Απορρίπτεται. 96. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται 97. 7 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 98 υπέρ. Κατά αποχές. Η 98 απορρίπτεται. Η 8 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε, μάλιστα κυρία Ρεβονταλόν, νομίζω ότι η προσθήκη στην βιβαστική 7 υπήρχε κάποιος ο οποίος πραγματικά ήταν παρόν και δεν μπορούσε να ψηφίσει. Για μας είναι key vote, είναι καθοριστική και θα θέλαμε πραγματικά αυτό να επαναληφθεί, αυτή η συγκεκριμένη ψηφοφορία, αλλιώς στην τελική ψηφοφορία θα ψηφίσουμε αντίστοιχως. Μήπως θα μπορούσατε να σταματήσετε τις κατηδίαν συζητήσεις. Η κυρία Άντερσεν. Θα μπορούσαμε ίσως να ξεκαθαρίσουμε ποιος είναι ο σαφής κανόνας. Αν κάποιος είναι παρόν και αν μπορεί να μετρήσει ή όχι μια τέτοια ψήφος. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Όταν η πρόεδρος πει τέλος της ψηφοφορίας, η ψηφοφορία έχει τελειώσει. Αυτός είναι ο κανόνας. Μάλιστα, έχετε το λόγο. Συγγνώμη, Πρόεδρε, αλλά και στην αίθουσα οι Πρόεδροι ρωτούν αν έχουν ψηφίσει όλοι και στην Ολομέλεια. Μισό λεπτό να βάλει ακουστικά η Πρόεδρος, γιατί δεν ακούω. Κύριο Σασόλ. Και στην αίθουσα της Ολομέλειας, κυρία Πρόεδρε, όταν ε, προεδρεύει κάποιος, ρωτά τους βουλευτές αν έχουν ψηφίσει όλοι. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα καλός τρόπος, διότι μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους κάποιο ε, δεν μπόρεσε να ψηφίσει, δεν πάτησε ένα κουμπί. και δεν κατάφερε να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου του. Το να ρωτήσουμε τους παρισταμένους εάν ψήφισαν όλοι, θεωρώ ότι είναι καλός κανόνας. Κοιτάξτε, δεν έχουμε πολύ ώρα να χάσουμε με το ίδιο θέμα. Θα σας δώσω το λόγο για ένα λεπτό γιατί πραγματικά έχουμε ήδη καθυστερήσει. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να σας υπονθυμίσω ότι ήταν η δεύτερη ψηφοφορία. Ήδη την έχουμε επαναλάβει μια φορά. Και ήταν σαφές αρχή της ψηφοφορίας, τέλος της ψηφοφορίας. Και μόνο όταν αποφασίσατε να ανακοινώσετε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Αποφάσισε τη σοσιαλιστική ομάδα ότι δεν μπόρεσε ένας ε, να ψηφίσει. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει το ίδιο τρεις, τέσσερις, πέντε φορές και να είχαν μπει ένα, δύο ή τρία άτομα. Δύο φορές έγινε η ίδια ψηφοφορία. Δεν νομίζω ότι πρέπει να το ξανακάνουμε άλλη μια τρίτη φορά. Νομίζω ότι ήμασταν αρκετά υπομονετικοί έχω την εντύπωση ότι πρέπει να παραμείνουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν είναι δυνατόν, σέβομαι τους συναδέλφους, αλλά πραγματικά δεν μπορεί να περιμένουμε ο καθένας που μπήκε καθυστερημένα να μπορεί να επαναλάβει την ψηφοφορία. Μάλιστα έχετε το λόγο. Και κατόπιν εσείς. Κοιτάξτε, Ξεκινάμε την ψηφοφορία στις 9. Το λέει ρητά και σας παρακαλώ πολύ, μπορείτε να είστε στην αρχή της ψηφοφορίας και όχι καθυστερημένοι 10 λεπτά. Κάποιοι είναι στην ώρα τους. Αν δεν είστε στην ώρα σας, τότε δεν μετράει η ψήφο σας. Είναι πολύ απλό. Σας παρακαλώ πολύ, μην χειροκροτείτε. Μπορεί κάποιος να καθυστερήσει, εντάξει. je suis bien και το ξέρω αυτό γιατί πολλές φορές ξέρετε ότι μου συμβαίνει και εμένα σε αντιπροσωπείες. Κυρία Φώστερ, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι επειδή είμαι το αρχαιότερο μέρος εδώ στην Επιτροπή, έχω την εντύπωση ότι το 1999 άλλαξαν οι κανόνες και είναι σαφέστατοι. Νομίζω ότι μπορεί όλοι να μπούμε σε μια ψηφοφορία είτε στην Ολομέλεια είτε στην Επιτροπή γιατί ήμασταν κάπου αλλού. Και πραγματικά πρέπει να είναι κάποιος καθιστός στη θέση του και να είναι έτοιμος να ψηφίσει. Νομίζω πραγματικά ότι πρέπει να είμαστε αυστηροί σε αυτό. Και όπως είπε και ο συνάδελφος, το συζητήσαμε επαναλάβαμε την ψηφοφορία και νομίζω Πρόεδρε, δώσατε αρκετό χρόνο στα άτομα που μπήκαν για να μπορέσουν να συμμετάσχουν. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι όλοι πρέπει να προσπαθούμε να είμαστε στην ώρα μας πριν ξεκινήσει μία ψηφοφορία και θα πρέπει από εδώ και πέρα να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ κυρία Φώστερ. Ποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο? Κυρία Κίλαναν, θέλετε το λόγο? Η κυρία Κίλανεν δεν θέλει ε, το λόγο, θέλει να τα πει όλα. Εντάξει, πέρα της ψηφοφορίες, αφού θέλετε αυτό να πω και δεν επανερχόμαστε. Αποφασίζω λοιπόν τώρα ότι ψηφίζουμε το σύνολο της έκθεσης. Άρχεται η ψηφοφορία, τελική ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. της Απορρίπτεται η έκθεση με μεγάλη πλειοψηφία. une Πρόκειται για γνωμοδότηση για έκθεση της Επιτροπής ΕΝΒΙ και ΙΤΡ. Ορίστε. Συνεχίζουμε λοιπόν τη συνεδρίασή μας. Αν θέλετε να βγείτε, να βγείτε ήσυχα, γιατί συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Συνεχίζουμε λοιπόν. Αγαπητοί συνάδελφοι, αν θέλετε να μιλήσετε, κάντε το έξω. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα έξυπνα συστήματα μεταφορών. Τα συνεργατικά συστήματα. Εισηγητή μα, ο κύριος Ούλριχ. Αυτό δεν γίνεται. Αν θέλετε να συζητάτε μεταξύ σας, βγαίνετε έξω. Ευχαριστώ. Allez, nous continuons. Συνεχίζουμε λοιπόν. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον εισηγητή μας και μετά θα συνεχίσουμε με τους κοιόδης. Κύριε Ουλρικ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους εμπειρογνώμονες και τις οργανώσεις εμπειρογνωμόνων που ήρθαν εδώ για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για αυτήν την έκθεση. Επίσης, να ευχαριστήσω τους επισκέπτες που έχουν έρθει εδώ από την Ουγγαρία. Μας τιμούν, μας τιμάει η περιέργειά τους. Έχουμε εδώ φοιτητές αλλά και συνταξιούχους από το κοινοβούλιο. Να μην το κάνετε αυτό γιατί αν χειροκροτείτε η πρόεδρος θα μας επιπλήξει. Βάλτε τις ζώνες σας γιατί θα μιλήσουμε για το μέλλον που γίνεται όλο και πιο γρήγορο. Επιταχύνουμε και είμαι σίγουρος ότι η κουλτούρα μας στις μεταφορές, τα οχήματα και τα πάντα θα αλλάξουν. Εδώ στην Επιτροπή Μεταφορών ασχολούμαστε με αυτό το θέμα πάνω από 10 χρόνια. Πώς θα φτιάξουμε έξυπνα συνεργατικά συστήματα μεταφορών και πώς θα τα εντάξουμε στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Σίγουρα θα έχετε δει την ταινία που έχουμε ε, έναν ε, οδηγό και τους επιβάτες που μπαίνουν στο αυτοκίνητο, πατάνε ένα κουμπί και ξεκινάει. Και αυτοί κάνουν τις, δουλειά, τις δουλειές τους. Όλα αυτά μοιάζουν με επιστημονική φαντασία και ότι δεν είναι πραγματικά ή ρεαλιστικά. Βέβαια η έκθεσή μου δεν είναι γι' αυτό το θέμα, αλλά στην ουσία θα... να τονίσω ότι ε, εμείς με αυτή την έκθεση προσπαθούμε να θέσουμε τη βάση για την εφαρμογή ενός συστήματος ε, το οποίο θα μπορέσει να επιβιώσει στην εποχή των συνεργατικών έξυπνων αυτοκινήτων. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου, ο Τίλα Μπένεντεκ και εσύ αξίζει χαρητήρια ήσουν μεταξύ αυτών που μας ε, βοήθησαν. Υπάρχουν όμως και άλλοι που πάνε από τις ΗΠΑ μέχρι την Κίνα, το Βερολίνο και άλλα μέρη και άλλες χώρες. Υπάρχουν πολλοί εμπειρογνώμονες και οργανώσεις που μα έδωσαν πληροφορίες σχετικά με το πώς θα είναι το μέλλον. Αυτό για το οποίο συζητάμε σήμερα είναι ένα σύστημα όπου τα ε, οχήματα συνεχώς επικοινωνούν μεταξύ τους. Αυτό θα βοηθήσει στην ασφάλεια, στην αποφυγή ατυχημάτων, διότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους λόγω ατυχημάτων, τροχαίων ατυχημάτων κάθε χρόνο. Συνεπώς η ασφάλεια και η προστασία αυτών των ανθρώπων είναι το πρώτο μας μέλημα. Σε πολύ λίγα χρόνια θα έχουμε εντελώς καινούργια αυτοκίνητα, εντελώς καινούργια οχήματα στους δρόμους μας. Θα επικοινωνούν μεταξύ τους μέσα από μηχανήματα, οδικά συστήματα που θα τους φέρνουν σε επαφή, θα τα φέρνουμε σε επαφή με τα κέντρα ελέγχου κυκλοφορίας σε 24 ώρες το 24ωρο, όποτε βγαίνουν στο δρόμο για να πάνε κάπου. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν. Μπορούμε να αποφύγουμε ανθρώπινα λάθη, να λάβουμε υπόψη μας τις μετεωρολογικές συνθήκες αν υπάρχει ατύχημα. Το σύστημα μπορεί να στείλει άμεσα πληροφορίες ε, για την ακριβή τοποθεσία στην οποία συνέβη το ατύχημα ε, στο ΕΚΑΒ, ε, στα, στις άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Αν υπάρχει κάποια βλάβη μπορεί να έρθει αμέσως η οδική βοήθεια. Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν πρέπει να ε, μείνουμε πίσω από τις εξελίξεις, γιατί είμαστε πραγματικά πίσω σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα που ακολουθεί. Θα θέλαμε λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το σύστημα να εισαχθεί άμεσα. Πώς θα γίνει αυτό όμως όταν ακόμα και ανάμεσα στα κράτη-μέλη υπάρχει μεγάλο χάσμα σε επίπεδο εξέλιξης. Θα σας μιλήσω για τη χώρα μου, την Ουγγαρία. Προφανώς δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το κέντρο της Βουδαπέστης και το επίπεδο εξέλιξης εκεί και με μία ε, πόλη, έναν οικισμό 150 χιλιόμετρα μακριά. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές και αυτό ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη. Αγαπητοί συνάδελφοι, λοιπόν, αυτή η έκθεση είναι ε, μια καυτή πατάτα, ένα ζεστό ε, καυτό ζήτημα. Ε, όλοι ενδιαφέρονται γι' αυτό. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες, οι πάντες. Πρέπει λοιπόν αργά ή γρήγορα να αποφασίσουμε σε ποια κατεύθυνση θα πάμε. Να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί πάντοτε είναι διαθέσιμη. Εγώ ως εκπρόσωπος της Επιτροπής μας και υπεύθυνο για αυτό το θέμα έχω λάβει ε, μεγάλη ε, βοήθεια από τη Γενική Διεύθυνση MOVE MV ε, και τους ευχαριστώ όλους για τη δουλειά τους. Επίσης υπάρχουν δύο ε, ομάδες εμπειρογνωμόνων. Η πλατφόρμα ITS ήταν μία από αυτές τις οργανώσεις και μας βοήθησε να συνοψίσουμε τη δουλειά 8 ε, ομάδων εμπειρογνωμόνων. Το 2021 θα είναι το έτος ε, της ηλεκτροδότησης, της συνδεσιμότητας, το ε, έτος της αυτοματοποίησης και των ηλεκτρικών οχημάτων. Εμείς θέλουμε να συνδέσουμε τις τηλεπικοινωνίες με την αυτοκινητοβιομηχανία, τις μεταφορές, της τεχνολογίας των πληροφοριών. Όλοι αυτοί οι κλάδοι πρέπει να συνεργάζονται για να μπορούμε να εισαγάγουμε αυτό το σύστημα και να υιοθετήσουμε και τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Πολύ σημαντική λοιπόν η συνεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και μεταξύ των κρατών μελών. Ή δυνατόν όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μπουν στο πρόγραμμα Sea Roads. Α, εφόσον έχουμε σπαταλήσει τόσο χρόνο με την ψηφοφορία, δεν θα μπορέσω τώρα να μπω στις λεπτομέρειες, γιατί η έκθεση είναι μακροσκελής. Υπάρχει όμως ένα θέμα που θέλω να αναφέρω. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές που περιμένω σε σχέση με την ανακοίνωση της Κομισιόν, Συμφωνώ πλήρω ε, με την ε, κατεύθυνση της Κομισιόν ως μέλος των σοσιαλιστών. Δεν μπορώ ε, να το πω πιο δυνατά. Δεν μπορώ να δώσω μεγαλύτερη έμφαση. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι όποιο σύστημα εισάγουμε, εισαγάγουμε θα πρέπει να έχει σε αυτό πρόσβαση ο καθένας πολίτης δεν μπορούμε να το έχουμε διαθέσιμο μόνο για τους πολίτες των πλούσιων χωρών. Πρέπει να φτάσουμε στον απλό πολίτη, στον κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι πρέπει να υποφεληθούν από αυτό το νέο σύστημα και τη νέα αυτή επανάσταση. Γιατί η ζωή αυτών των ανθρώπων αξίζει το ίδιο με τη ζωή των πλουσίων που ζουν στις πόλεις. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε την ίδια ε, προστασία, το ίδιο επίπεδο προστασία σε όλους τους πολίτες όσον αφορά στα ατυχήματα. Μίλησα για τη βιασιμότητα, τη συνδεσιμότητα ε, ως προτεραιότητες. Να ευχαριστήσω την Πρόεδρο, διότι πραγματικά έχουμε δώσει μια πράσινη προσέγγιση σε αυτή την έκθεση. Είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε και για το περιβάλλον, για το φόρτο για το πόσο επιβαρύνεται το περιβάλλον. Επίσης, χρειαζόμαστε την κυβερνοασφάλεια και την προστασία ε, του κυβερνοχώρου και των δεδομένων. Γιατί φανταστείτε την ποσότητα των δεδομένων, τον όγκο των δεδομένων που ανταλλάσσονται μέσα από αυτά τα συστήματα των έξυπνων οχημάτων. Υπάρχουν τρίτοι οι οποίοι μπορούν να ε, υποκλέψουν τα στοιχεία αυτά, να χακάρουν ε, και να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία για εμπορικού ε, σκοπούς και άλλους σκοπούς. Να τονίσω ότι στην παράγραφο 15 αναφέρεται το ETSI και το σύστημα ETSG5 και τα συστήματα των εφαρμογών για κινητά που ήδη υφίστανται. Και έχω και, στα, και μέσα στις παρενθέσεις ε, τα μελλοντικά δίκτυα. Ε, θα κάνω κάποιες αλλαγές λοιπόν με βάση τόσα μου είπαν οι εμπειρογνώμονες πρόσφατα. Θέλουμε αυτές οι τεχνολογίες να επικοινωνούν μεταξύ τους. Και άλλη μια παράγραφος ε, είναι η 20 η οποία πάει πέρα από το CITS πέρα δηλαδή από τα συνεργατικά έξυπνα συστήματα μεταφορών. Ε, δυστυχώς εδώ δεν υπήρξε λύση ε, που να αποδέχονται όλα τα μέρη. Ε, μιλάμε για ένα νομοθετικό πλαίσιο που να καλύπτει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να δημιουργεί την διαλειτουργικότητα που χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε λοιπόν νομοθεσία η οποία θα δημιουργεί ίσους όρους και συνθήκες για πρόσβαση στα έξυπνα οχήματα. Την ίδια στιγμή όμως πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας την ε, καινοτομία, τον ε, θεμητό ανταγωνισμό και την ίση μεταχείριση των πολιτών. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχω ε, στο μυαλό μου και αυτά προσπαθήσαμε να βάλουμε και στις τροπολογίες. Για παράδειγμα, αστικές μεταφορές. πεζοί, ποδηλάτες, μοτοσικλετιστές. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ευάλωτοι, είναι οι ευαίσθητες ομάδες ε, του συστήματος μεταφορών. Ευχαριστώ τους συναδέλφους λοιπόν από την Κομισιόν ε, και από το Κοινοβούλιο. Ε, για την δουλειά που επέρχεται. Είμαι έτοιμος να δεχτώ ένα τσουνάμι από τραπολογίες και θα χαρώ γιατί αυτό θα δείξει ότι όλοι θέλουν να ασχοληθούν με το θέμα. Ευχαριστούμε τον κύριο ε, Πριν ξεκινήσει η συζήτηση, ε, να έλθω λίγο στους επισκέπτες μας. Έχουμε μέλη από το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, είναι συνταξιούχοι ε, από το Σύλλογο των Συνταξιούχων του Κοινοβουλίου και εκπροσωπούν γενικά τους συνταξιούχους από την Ουγγαρία. Ε, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Ξεκινά αμέσως η συζήτηση. Ξεκινάμε με σας, κυρία Έρκινεν. Έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ τον εισηγητή για την παρουσίαση και το σχέδιο έκθεσης. Συμφωνώ ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Όπως ξέρουμε, η αυτοκινητοβιομηχανία είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Ευρώπης. Είναι σημαντικό να ηγούμαστε και σε αυτό το τομέα. Ξέρουμε ότι στις ΗΠΑ και την Κίνα υπάρχουν τεράστιες εξελίξεις Υπάρχουν συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούν πλέον. Πρέπει λοιπόν και εμείς να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Γιατί αυτή η βιομηχανία είναι μία από τις βασικέ βιομηχανίες που συνεισφέρει στον προϋπολογισμό μας. Ε, ε, θα πρέπει λοιπόν να αναπτύξει και αυτή δράση για την ψηφιοποίηση, να έχουμε ε, λοιπόν κάθε δυνατότητα να επιτρέψουμε στη βιομηχανία αυτή να ευημερίσει περαιτέρω σε επιχειρησιακή βάση. Αυτή η εκθέση είναι πολύ καλή για τη μελλοντική δουλειά που θα γίνει. Τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής είναι ευπρόσδεκτα, τα χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε τα έξυπνα συνεργατικά συστήματα μεταφορών και τα αντίστοιχα οχήματα. Θέλουμε πιο ασφαλείς δρόμους και πιο καθαρό περιβάλλον. Αυτά όλα τα βλέπουμε εδώ. Αν μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την ψηφιοποίηση, την ψηφιακή τεχνολογία, θα έχουμε πιο βιώσιμα και πιο αποτελεσματικά συστήματα μεταφορών. Κάτι που χρειαζόμαστε πολύ, διότι ξέρουμε ότι ο αριθμός των οχημάτων συνεχώς αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη. Απαιτούνται λοιπόν νέες λύσεις. Επίσης θεωρώ ότι η δική μας έκθεση πρέπει να είναι λίγο πιο φιλόδοξη. Θα ήθελα να ε, δω και κάποιους πιο συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα. Πώς θα επιτύχουμε αυτά τα σημαντικά ε, βήματα τα επόμενα ε, χρόνια. Επίσης είμαι υπέρ της υβριδικής προσέγγισης, ας πούμε συμπληρωματικές τεχνολογίες πληροφοριών. Αυτό καλύπτεται νομίζω. Ε, πρέπει να είναι αξιόπιστες αυτές οι συνδέσεις. Αυτό πρέπει να μπορούμε να το εγγυηθούμε. Και κάτι άλλο που ήδη υπογράμμισε ο εισηγητής είναι ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που χρειάζεται να τα σκεφτούμε καλά η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η προστασία των δεδομένων. Όπως ξέρετε, η ιδιωτικότητα και η προστασία των ε, προσωπικών δεδομένων είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία. Οι χρήστες πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν τα δεδομένα τους. Ταυτόχρονα να υπογραμμίσω και εγώ αυτό που είπε ο εισηγητής. Η παράγραφος 20. πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να διασφαλίσουμε ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και τους σπόρους ε, για τα οχήματα, γιατί χρειάζεται καινοτομία εκεί και πρέπει να βρούμε και τους σπόρους για αυτήν. Αν θέλουμε καινοτόμα προϊόντα, χρειαζόμαστε προστασία ε, αλλά και πρόσβαση στα δεδομένα που, ε, που δίνουν αυτά τα οχήματα. Επίσης ε, πρέπει να έχουμε και χρηματοδότηση για πιλωτικά προγράμματα. Η Κομισιόν πρέπει να διασφαλίσει ότι η αυτοκινητοβιομηχανία θα παραμείνει πιστή στην δέσμευσή της να ε, ξεκινήσει την πλήρη εφαρμογή αυτών των οχημάτων, οχημάτων μέχρι το 2019. Χρειαζόμαστε λοιπόν να αξιολογήσουμε προσεκτικά τους κανονισμούς ε, που διέπουν αυτόν τον τομέα. Να μην ε, ρυθμίζουμε υπερβολικά. Να αφήνουμε περιθώριο για την καινοτομία. Το πιο σημαντικό όμως είναι να υποστηρίξουμε μία προσέγγιση η οποία θα δημιουργήσει ένα πλαίσιο φιλικό προς την καινοτομία. Να ε, υπογραμμίσω επίσης και την ανάγκη να υπάρχουν ενημερωμένες εθνικές νομοθεσίες για αυτό τον τομέα σε πολλά κράτη-μέλη ίσως η νομοθεσία να μην είναι ενημερωμένη, να μην είναι φιλική προς, τις, την καινοτομία. Άρα θα πρέπει να ενθαρρύνουμε και τα κράτη-μέλη με τη σειρά τους, όπως και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι, να κάνουν αυτό που χρειάζεται, γιατί είναι μια κοινή προσπάθεια. Καλό λοιπόν και τον εισηγητή και όλους τους συναδέλφους από την πλευρά της Επιτροπής Μεταφορών να έχουμε μια φιλόδοξη στρατηγική. Δυστυχώς πρέπει να προλάβω την πτήση μου και δεν, πρέπει, δεν μπορώ να μείνω για όλη τη συζήτηση, αλλά οι συνάδελφοι εδώ που είναι ιδιαίτερα ενεργοί στο θέμα θα συμμετάσχουν σε όλη τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Δέμεσμέκερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν είμαι σκιώδης εισηγητής, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό, πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση ε, και να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για την πολύ καλή προσέγγιση. Είμαι βέβαιος ότι εδώ στο Κοινοβούλιο θα δοθεί ένα πολύ ε, ισχυρό μήνυμα ότι είμαστε πρωτοπόροι για τις ε, συνεργατικές συνδεσμένες ε, μεταφορές. Ε, τα συστήματα CITS μπορούν να εξασφαλίσουν ασφάλεια, άνεση στην οδήγηση, αλλά μακροπρόθεσμα νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και τι δυνατότητες έχουν αυτά τα συστήματα να λειτουργήσουν στις συνδυασμένες μεταφορές. Ο εισηγητής πολύ σωστά αναφέρθηκε στη διαλειτουργικότητα, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διαλειτουργικότητα των διαφόρων συστημάτων. Πιστεύω ότι χρειάζεται ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα παρέχει και ασφάλεια δικαίου ε, ώστε στη συνέχεια να προωθήσουμε και τις επενδύσεις. Επίσης θα ήθελα να επισημαίνω ότι η αυτοκινητοβιομηχανία είναι διεθνής εκφύσεως. Θα πρέπει να ε, συνομιλούμε με τους πιο σημαντικού μας εμπορικούς εταίρους, ώστε να είναι όσο πιο δίκαιες οι συνθήκες γίνεται. Έχω και κάποια ακόμα σχόλια και θα υποβάλω σχετικές τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντεμεσμάκερ. Ο κύριος Βαν Μίλτονμπερκ έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα συνεχίσω στα αγγλικά. Καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και να ευχαριστήσω τον εισηγητή για ε, πραγματικά ε, ένα εξαιρετικό σχέδιο έκθεσης, το οποίο σαφέστατα καθορίζει δικαιώματα και προτεραιότητες και συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει να τονίσουμε την ε, προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ιδιωτική ζωή, την κυβερνοασφάλεια και αυτά συνάδουν με το σχέδιο έκθεσης του εισηγητή, ο οποίος σε μία δήλωση ε, λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ε, θεσπίσει ταχύτητα ένα κατάλληλο πλαίσιο ώστε να ξεκινήσει η διαλειτουργικότητα όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 27. Συμφωνώ απολύτως λοιπόν με αυτό και εδώ θα πρέπει να επιδείξουμε και τη δέωσα φιλοδοξία. Θεωρώ επίσης ότι το CITS ε, θα συμβάλλει ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές και πιο βιώσιμες οι οδικές μεταφορές και είναι λογικό να υπάρχουν όλο ένα και περισσότερες λύσεις CITS ε, στα οχήματα. Αναφέρθηκε άλλωστε και στι ε, παρεμβάσει των ε, προηγούμενων συναδέλφων. Και όπως και οι υπόλοιπες ομάδες υποστηρίζω μια φιλελεύθερη προοπτική της αγοράς. Πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερη αυτή η πρόταση. Ε, ούτως ή άλλω, του κανόνε θα του καθορίσει τελικά η αγορά και η αγορά θα μα δώσει και τις λύσεις που χρειάζονται. Όμω, η ασφάλεια των χρηστών και των πολιτών είναι πάρα πολύ σημαντική για μας ε, ω ομάδα των φιλελευθέρων, Επομένω, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα οχήματα τουλάχιστον μακροπρόθεσμα, τουλάχιστον μακροπρόθεσμα θα επικοινωνούν μεταξύ του. Ε, στη μεταβατική περίοδο θα πρέπει να σκεφτούμε πώ μπορούμε να έχουμε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ οχημάτων που φέρουν και οχημάτων που δεν διαθέτουν τη δυνατότητα διασύνδεσης. Ε, και υπάρχει και η ε, λεγόμενη ε, συμβατότητα ε, προς το πιο αρχαίο, προς το πιο παλιό. Και εδώ ζητώ να ληφθούν υπόψη τα δικαιώματα των καταναλωτών ως προς την ιδιωτική του ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα και θα ήθελα να ζητήσω να υπάρχει κατάλληλη εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων από πλευρά Επιτροπή. Επιπλέον, οι κατασκευαστέ ποτέ δεν θα πρέπει να κάνουν επεξεργασία των δεδομένων εντό του οχήματο χωρί να υπάρχει ρητή συγκατάθεση ε, του χρήστη ή του οδηγού του αυτοκινήτου ε, και ελπίζω να περάσουν και αυτό στην του CITS και να αναφέρεται και στο σχέδιο έκθεση του εισηγητή. Επίσης, θα ήθελα να ζητήσω να υποστηρίξουμε την παρούσα ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, για παράδειγμα μέσω της πλατφόρμας CATS και θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρχει ε, υπάρχουν ε, ε και ε, εθνικοί ε, πυλώνες του CITS που χρειάζονται και την κατάλληλη υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θεωρώ, κύριε Πρόεδρε, για να ολοκληρώσω, ότι όλα αυτά τα οποία προτείνει ο Συγητή, συνάδουν με τι απόψει μου ω ισχυώδη εισηγητή. Θα προτείνω λοιπόν ελάχιστε τροπολογίε που αφορούν κυρίω ε, ε, καταναλωτικό δίκαιο και ε, ουδετερότητα σε τεχνολογικό επίπεδο. Θα υπάρχει όμως μια συγκεκριμένη τροπολογία στην παράγραφο 21 για το διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους. Ε, Καταλαβαίνω ο εισηγητή είναι σοσιαλιστή και δημοκράτη. Ε, θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν παράγραφο για τον κοινωνικό διάλογο, την οποία επικροτώ, αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι το CITS ε, αφορά και την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των θετικών και των αρνητικών συνεπειών που θα μπορούσε να έχει ε, σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο, ε, διότι θα δημιουργήσει θέσει εργασία, θα δώσει όθηση στην οικονομική ανάπτυξη και θα υπάρχουν φυσικά και κάποια άλλοι τομεί οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν ε, προβλήματα και δεν θα μπορέσουν να διαφυλάξουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας. Εμείς θα πρέπει όμως να έχουμε μια θετική στάση, να υπάρχει μια αισιοδοξία ε, προς την πρόοδο, αυτό το υποστηρίζει και η ομάδα μου και ελπίζω να συνεργαστούμε με τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές για ένα πολύ συναρπαστικό θέμα και είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να επιδείξουμε την ίδια συνεργασία ε, στην κοινή μας προσέγγιση όπως αναφέρεται και στον τίτλο του κειμένου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Βαν Μίλτενμπεργκ. Η κυρία Κίλων έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το πρώτο και το κυριότερο είναι ο νέος ε, τρόπος σκέψης, η νέα νοοτροπία. Να δούμε αυτά τα οχήματα με μια νέα προοπτική και να έχουμε υπόψη μας ε, τις υπηρεσίες σε όλες τις μεταφορές. Να δώσουμε όθηση στις συνδυασμένες μεταφορές με το CITS και νομίζω ότι η προσέγγιση που θα ε, έχει στο επίκεντρο τον πελάτη είναι ε, η πλέον απαραίτητη. Η έκθεσή σας κύριε Σιγητά αποτελεί πολύ καλό υπόβαθρο για να ξεκινήσουμε τις περαιτέρω συζητήσεις μας για το θέμα αυτό και πιστεύω ότι θα πρέπει να ξεκινήσει ο διάλογος ε, με τους πελάτες. Τι ανάγκες έχουν, τι ελπίδες έχουν οι πελάτες, ε, οι επιχειρήσεις, ε, ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες ε, να υπάρχει ρύθμιση στον τομέα αυτό και τι δεν χρειάζεται να ρυθμίσουμε, αλλά και πού υπάρχει ανάγκη να δώσουμε όθηση, για παράδειγμα, με μέσα χρηματοδότησης. Πιστεύω ότι το ITS ε, σχετίζεται άμεσα με τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών, την ενιαία, μεταχωρά, την ενιαία αγορά και την ενεργειακή ένωση. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Και φυσικά όλα αυτά μας συνδέουν και ε, με θέματα διασυνοριακής ε, συνεργασίας, την οποία χρειαζόμαστε κατεπηγόντως. Το σύστημα ITS ε, θα μας βοηθήσει να διορθώσουμε τα ανθρώπινα σφάλματα και τις άλλες ατέλειες των συστημάτων που έχουμε αυτή τη στιγμή, αλλά και ό,τι άλλο σχεδιάζουμε στο μέλλον και θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε. σε θέματα ασφάλειας και προστασίας ή κυβερνοασφάλειας ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας και αυτή τη συνεργασία μεταξύ των οχημάτων και να υπάρχουν και κατάλληλες τεχνολογίες και σχετικά επιχειρηματικά μοντέλα στις οδικές μεταφορές. Υπάρχει η σύνδεση, αλλά ακόμα δεν συνεργαζόμαστε αρκετά και νομίζω ότι το CITS θα μπορούσε να αποτελέσει λύση. Να υπάρχει διασύνδεση, αυτοματοποίηση, ε, να υπάρχει ευφυής χρήση ε, των καυσίμων, κατάλληλη ενεργειακή κατανάλωση, μπορεί να δώσει όθηση στην ανταγωνιστικότητα σε όλη την Ευρώπη, αλλά πιστεύω ότι χρειαζόμαστε επίσης και κατάλληλη χρηματοδότηση και επιδοτήσει σε όλους τους τομείς και με αυτόν τον νέο τρόπο, να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε όλα τα κράτη-μέλη για περιφερειακή ανάπτυξη των πόλεων, ε, υπάρχουν διάφορες ανάγκες και πρέπει να εξασφαλίσουμε και ότι το CITS θα μας επιτρέψει να έχουμε διασύνδεση και να έχουμε και πλήρη συμμόρφωση και ε, πλήρη απεξάρτηση από τον άνθρακα. Θεωρώ ότι αυτά αποτελούν τη ραχοκοκαλιά και είναι επίγον να συνδεθούν οι Ευρωπαίοι με αυτές τις νέες ιδέες και το νέο σκεπτικό. Προς το παρόν η ανάπτυξη είχε ως κύριο μοχλό την ε, τεχνολογία. Χρειαζόμαστε κατεπηγόντων μελέτες ε, και να αναγνωρίσουμε και την ε, ανθρώπινη πτυχή και την κοινωνική πτυχή αυτών των θεμάτων και να εξασφαλίσουμε ότι θα λάβουμε υπόψη μας τις περιβαλλοντικές, τις κοινωνικές και τις ανθρώπινες αξίες. Να μην δούμε μόνο την τεχνολογική σκοπιά. Και κάτι τελευταίο, Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό δίδαγμα που μάθαμε από τη Silicon Valley στην Καλιφόρνια είναι το εξής μήνυμα. Αυτοί που λένε ότι δεν μπορεί να γίνει, δεν θα πρέπει να ανακόψουν την πορεία αυτών που το υλοποιούν. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια εξαιρετική συμβουλή προς τους ηθήνοντες. Και με αυτό θα ολοκληρώσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Προσβλέπω στη συνεργασία και με πολύ μεγάλη αγάπη. Ευχαριστώ κύριε Κιλώνεν. Ο κύριο Δενταλούντε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για ένα πολύ καλό σχέδιο κειμένου. Θα θέλαμε να τονίσουμε τρία πράγματα. Πρώτον, υποστηρίζουμε ακράδαντα την παράγραφο 12 για την ιδιωτική ζωή και την προστασία δεδομένων και την παράγραφο 14 για την κυβερνοασφάλεια, που θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικέ. Θα θέλαμε όμως να υπάρχει και πιο ισχυρή διατύπωση ακόμα για να υπάρχει καλύτερη συντονισμό και συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να αναφερθούμε και στην ε, Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών για την προσβασιμότητα για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα για να υπάρχει πλήρης πρόσβαση στο CITS ε, για όλου του πολίτε. Τρίτον, για την παράγραφο 19 για τι συνδυασμένε μεταφορέ. Νομίζω ότι οι κρατήσεις ε, εισιτηρίων και η έκδοση εισιτηρίων θα πρέπει να συμπεριληφθούν εδώ για να έχουμε πόρτα-πόρτα ε, όλα αυτά τα πράγματα και εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να αναφερθεί και η ποδηλασία. Ευχαριστώ κύριε Νταλούντε. Η κυρία Αρνοτσού. Δεν θέλει το λόγο. Ο κύριος Λόγκριν επίσης δεν θέλει το λόγο. Θέλετε το λόγο. Παρακαλώ. Με ξέρετε, εμένα μου αρέσουν τα αυτοκίνητα, έχω 9 οχήματα και έχω και δύο ε, αυτοκίνητα αγώνων και έχω και ηλεκτρικό όχημα. Υπάρχει όμως ένα όχημα το οποίο ποτέ δεν θα καταλήξει στον καράς μου και είναι αυτό το οποίο δεν μπορώ να το οδηγήσω γιατί μου αρέσει η οδήγηση και δεν θέλω να είμαι απλώς επιβάτης ε, στο αυτοκίνητό μου και ε, θέλω να είμαι εγώ αυτός ο οποίος αποφασίζει για το αυτοκίνητο. Ε, και νομίζω ότι είμαι αρκετά μεγάλο πλέον, είμαι 54 ετών και ελπίζω ότι θα έχω πεθάνει πριν έρθει η επανάσταση των οχημάτων χωρί οδηγό που θα εμφανιστούν στου δρόμου. Θα απολαύσω λοιπόν το τελευταίο τμήμα της ζωής μας τρέχοντας, χρησιμοποιώντας ε, τι αντίκε μου και τα αυτοκίνητά μου και να απολαύσω μια ζωή που θα αγαπώ ε, το αυτοκίνητο. Κύριε Λούντκριν, μπορεί και να σας εκπλήξει η τεχνολογία γιατί προχωρά τόσο γρήγορα που ακόμα και εσείς, ε, κύριε Λάνγκριν κύριε Λάνγκριν σας μιλάω. Κύριε Λάνγκριν λοιπόν, αν αγαπάτε λοιπόν το αυτοκίνητο, θα αγαπάτε και αύριο το αυτοκίνητο, κύριε Λάγκριν. Θα είναι πιο καθαρό, θα είναι συνδεδεμένο και εσείς δεν θα έχετε τίποτα να κάνετε. Ε, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Και θα το λάβετε υπόψη σας γιατί θα είναι και κοινό το όχημα. Θα υπάρχει ε, μια συνεργασία. Ο κύριος Κόρ για ένα λεπτό γιατί καθυστερήσαμε πολύ στη συζήτηση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Ούνλικ για την πολύ καλή έκθεση. Ε, πρόκειται για μια καλή προσθήκη στη δική μου εκθεσή που θα ψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια. Νομίζω ότι και οι δύο εκθέσεις ακολουθούν την ίδια στρατηγική περισσότερη προστασία και ασφάλεια για τους καταναλωτές και όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο τους πλούσιους. Ε, θα ήθελα όμως ε, τώρα να μιλήσω για τα έξυπνα συστήματα πληροφορικής και επικοινωνίας όπως απαιτεί και η έκθεση. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα καλό βήμα προς την κατεύθυνση της υψηλής αυτοματοποίησης και με χαρά μου θα καταθέσω τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Μπάχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σημεία. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ τους συναδέλφους γιατί υπάρχει μια πολύ καλή βάση για συζήτηση και επεξεργασία. Υπάρχουν πολύ καλές προτάσεις, οι οποίες θα μπορούν να ενισχυθούν περαιτέρω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τις ε, διαφορές που υπάρχουν μεταξύ κάποιων ε, συγκεκριμένων προθεσμιών, μεταξύ των υποδομών που πρέπει να ολοκληρωθούν πριν ε, ξεκινήσει η παραγωγή κάποιων ε, αυτοκίνητων συγκεκριμένα. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα δεδομένα, όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα και ότι βεβαίως δεν θα πρέπει να είναι προσωπικά δεδομένα, δηλαδή να είναι δεδομένα τα οποία αναφέρονται σε συγκεκριμένα άτομα. Είναι πολύ σημαντικό εδώ να αγγιθούμε με νέα συστήματα ασφαλείας και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και να μην, αν θέλετε, περιοριστούμε μόνο στο θέμα της ε, μεταφοράς. Συγχαίρω τις προτάσεις των εισηγητών και όλη τους την προσπάθεια να ενσωματώσουν τις συνδυασμένες μεταφορές και βεβαίως ε, το γεγονός ότι θα υπάρχει πρόσβαση και θα είναι συνδεδεμένες όλες αυτές οι μεταφορές είναι το σημαντικότερο σημείο. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα. Καταλαβαίνω ότι είναι ευχάριστο για κάποιον οδηγεί όταν αγαπάει την οδήγηση. Εγώ είμαι φιλελεύθερη και φυσικά καταλαβαίνω ότι και αυτό θα πρέπει να το δεχτούμε. Από την άλλη, είναι πολύ σημαντική η ευκαιρία που μας δίνεται να αναπτύξουμε τις ε, συνδυασμένες μεταφορές και νομίζω ότι και ένας ε, οδηγός που του αρέσει η οδήγηση μπορεί να υποφεληθεί από αυτό γιατί θα είναι πολύ πιο ομαλή η κατάσταση. Στους δρόμους, παραδείγματος, θα υπάρχει περισσότερη ασφάλεια. Θα πρέπει λοιπόν να το δούμε σαν μια ευκαιρία. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Θα πρέπει να ενισχύσουμε μια πτυχή της έκθεσης αυτής, το θέμα της καθαρής ενέργειας, δηλαδή η συνθήκη του Παρισιού, οι δεσμεύσεις της ΚΑΠ 21, αναφέρουν στην ε, ποιότητα του αέρα και της ατμόσφαιρας στην Ευρώπη με ένα τεράστιο ακόμα αριθμό θανάτων που οφείλεται στην μόλυνση. Επίσης το θέμα της ε, κινητικότητας η οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και πολλούς άλλους τομείς. Σήμερα στην Ευρώπη βλέπουμε ότι το 13% του προϋπολογισμού των νοικοκυριών διατίθεται για τις μεταφορές. Αυτό είναι ήδη ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Την ίδια ώρα βλέπουμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ κάποιων περιοχών και κάποιων άλλων. Αυτό το διαπιστώνουμε σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Μεταξύ αστικών περιοχών και υπαίθρου. Μεταξύ γενεών. Ο ψηφιακό κόσμος μας ε, έδειξε την κατάφορη αδικία και διαφορά που υπάρχει μεταξύ των κοινών. Όλοι οι νέοι έχουν ένα smartphone. Όμως όλοι δεν έχουν smartphone. Η κάλυψη επίσης ε, από το διαδίκτυο και αυτή δεν είναι ίση και δίκαιη. Ξέρουμε ότι θα περάσουν πολλά χρόνια μέχρι να επικρατήσει η ίδια ψηφιακή κάλυψη παντού στην Ευρώπη. Το θέμα των προσωπικών δεδομένων, ποιος θα έχει πρόσβαση, ποιος ε, θα τα διαθέτει, το θέμα της ασφάλειας του κυβερνοχώρου και το θέμα της αρμοδιότητας και της ευθύνης. Παραδείγματο χάρη δύο αυτόνομα αυτοκίνητα μπορεί ε, να έχουν ένα ατύχημα, ποιος είναι υπεύθυνος, ποιος έχει την αστική ευθύνη, η αυτοκινητοβιομηχανία, η κοινότητα η οποία δεν παρήχε σωστά δεδομένα. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα θέματα της αστικής ευθύνης, ας πούμε, είναι ένας τεράστιος τομέας ο θα πρέπει να ρυθμιστεί. Έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα τεχνικό θέμα και θα ήθελα να προσθέσω κάποια σημεία. Ευχαριστώ πολύ τους εισηγητές. Είναι εξαιρετική η έκθεση και μας προβάλλει στο μέλλον. Αυτά που ακούμε πολλές φορές πρέπει να τα φανταστούμε. Το θέμα όμως είναι ότι εργαζόμαστε με τα σημερινά δεδομένα και ο συνάδελφος Κοχ μίλησε για το θέμα της ηλεκτρονικής ε, στήριξης και ότι σήμερα μπορούμε να κάνουμε πιο ασφαλείς τις μεταφορές με τα συστήματα που υπάρχουν και τα οποία σήμερα υπάρχουν και λειτουργούν αυτόνομα στα αυτοκίνητά μας μία βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών που θα βασίζεται σε αυτά τα νέα συστήματα, στην τηλεματική παραδείγματος χάρη και το κατά πόσον η ακρίβειά τους μπορεί να βελτιωθεί και βελτιώνεται. Καλά, ο καθένας από εμά μπορεί να μιλήσει λέγοντας ότι ήδη στην Ασία η πρόοδος που έχει επιτευχθεί είναι τεράστια σε σχέση με την Ευρώπη και ότι τα συστήματα πλοήγησης των Αμερικανών είναι εξαιρετικά προηγμένα. Η ερώτηση που κάνω εγώ στην Επιτροπή τώρα είναι τι ακριβώς κάνουμε στην Ευρώπη, τα δορυφορικά συστήματα, το Γαλιλαίο. Αυτό είναι πιο σημαντικό για μένα από τις ακριβείς αποστάσεις που σήμερα προσπαθούμε να ρυθμίσουμε. Η ερώτηση για μένα είναι πόσο καλή ενεργειακή απόδοση μπορούμε να έχουμε και όχι μόνο το θέμα των συστημάτων ε, ε, πέδησης παραδείγματος χάρη και το πώς θα μεταβάλλεται η μικρή ενέργεια σε θερμότητα και θα ξαναχρησιμοποιείται από το κύκλωμα του αυτοκίνητου. Θέλω να πω, υπάρχουν γενικές ε, τεχνολογίες οι οποίες πρέπει καταρχήν να επιλεγούν ή να μην επιλεγούν και μετά θα δούμε τα επιμέρους θέματα που απορρέουν πρόσβαση στα δεδομένα κτλ. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια στον εισηγητή. Κοιτώ την DG Move. Θα σας δώσω το λόγο, αλλά σας παρακαλώ πολύ να είστε πάρα πολύ σύντομος. Α, κυρία Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος, γιατί όλα όσα άκουσα από την αρχή της συζήτησης το πρωί είναι πράγματα που αποσαφηνίζουν κάτι που ήθελα να πω και που είπα στην αρχή. Εμάς μας ενισχύουν αυτά που ακούμε από εσάς. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που δίνει ιδιαίτερες προοπτικές για τους πολίτες της Ευρώπης. Το θέμα της ασφάλειας. 26.000 νεκροί στους δρόμους της Ευρώπης κάθε χρόνο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ένα δις ευρώ είναι οι απώλειες που οφείλονται στη συμφόρηση της κυκλοφορίας στους δρόμους. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Πιστεύουμε ότι τα νέα συστήματα μπορούν να μας βοηθήσουν έτσι ώστε να ξεπεράσουμε αυτά τα δύο πολύ σημαντικά θέματα που μόλις σας προανέφερα. Η στρατηγική μας σας έχει ήδη ανακοινωθεί τα τελευταία δύο χρόνια. Τι έχουμε κάνει όμως περαιτέρω. Το θέμα της αυτοματοποίησης της σύνδεσης των έξυπνων αυτοκινήτων. Αυτό είναι κάτι που έχει προοδεύσει σημαντικά η στρατηγική μας. Βεβαίως σήμερα στοχεύει το πρώτο στάδιο. Η κοινή χρήση των ε, οχημάτων αυτών. Η αυτοματοποίηση είναι το δεύτερο βήμα. Υπάρχουν ε, ήδη πρωτοβουλίες και βεβαίως έχουν δημοσιευθεί και οι εκθέσεις που διευκρινίζουν και τα διάφορα στοιχεία τα οποία μέχρι τώρα έχουμε εντοπίσει σαν δυσκολίες. Είναι πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για την αυτοματοποίηση να πούμε με ακρίβεια πόσο γρήγορα θα προοδεύσει η τεχνολογία στους τομείς αυτούς. Πρέπει να ξεκινήσουμε από το 2019, αυτός είναι ο στόχος μας και αυτός ο στόχος πρέπει να στηριχτεί και από την αυτοκινητοβιομηχανία αλλά και από τις δημόσιες αρχές. Και χρειάζεται βεβαίως συντονισμός. Η οικογένεια των ε, συνδεδεμένων ε, δρόμων Sea Roads γιορτάζει σήμερα την επέτειο από την ε, πρώτη της θέση σε λειτουργία. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό στην Επιτροπή είναι ότι συνδυάζουμε αυτές τις πρώτες πρωτοβουλίες με τις νέες τεχνολογίες. Στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες και θα προσπαθήσουμε να θέσουμε όλον αυτό τον εξοπλισμό στην διάθεση των πολιτών, να τον κάνουμε κοινό κτήμα των Ευρωπαίων πολιτών. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους εμπειρογνώμονες για θέματα προστασίας των δεδομένων, συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη για τις ε, διασυνοριακές ε, δοκιμές και φυσικά συνεχίζουμε και επεξεργαζόμαστε το κείμενο της οδηγίας που έχει σήμερα δύο στόχους. Διαλειτουργικότητα είναι ο πρώτος στόχος. Αυτό θα πρέπει πραγματικά να ξεπεράσει τα σύνορα και τις μάρκες και τις αυτοκινητοβιομηχανίες και δεύτερον να υπάρχει συμβατότητα. Και αυτό είναι για να διασφαλίσουμε την απόδοση των επενδύσεων. Ολοκληρώνω Λέγοντα ότι με μεγάλη χαρά θα λάβουμε υπόψη μας όλα όσα ακούσαμε σήμερα στη ζήτηση αυτή στην έκθεση. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει και η έκθεση της ομάδας της DigiGrow, έκθεση της ομάδας υψηλού επίπεδου, οι οποίοι θα παρουσιάσουν αυτή την έκθεση εδώ στην Επιτροπή μας. Θα οργανώσουμε μια ακρόαση. Θα ακούσουμε λοιπόν σε αυτήν την ακρόαση τους εμπειρογνώμονες για το GEAR 2020. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό, κυρία Ούλρικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μισό λεπτό χρειάζομαι, γιατί νομίζω ότι όλη η συζήτηση δείχνει ότι υπάρχει ευρεία στήριξη και ενδιαφέρον για την έκθεση αυτή. Περιμένω τις προτάσεις των πολιτικών ομάδων και έχω μεγάλο πάθος και θα συνεχίσω με αποφασιστικότητα την επεξεργασία των προτάσεων σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών είναι η 21η Νοεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Συνεχίζουμε με τις εργασίες μας και τώρα θα μιλήσουμε με την Task Force. Tax Force. Sur la taxation du tourisme par la Commission européenne et la DG Gros, vous êtes... Πού Dans notre commission. Et donc vous... nous... Καλώς ορίσατε στην Επιτροπή Μεταφορών και θα μας παρουσιάσετε τις εργασίες σας. Υπεύθυνο για αυτήν την Task Force για τον τουρισμό είναι ο κύριος Ούληρη. Και μάλιστα για την ε, Παγκόσμια ημέρα του τουρισμού οργανώθηκε ένα φόρουμ εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δυστυχώς έχουμε καθυστερήσει, γι' αυτό και θα σας παρακαλέσω να είστε σύντομοι a turizmus albizottsága, a Tourism Task Force elején mindig tájékoztatást. Η Task Force για τον τουρισμό. Όταν μιλάμε για την Task Force για τον τουρισμό, Συνήθως ε, δίνουμε πληροφορίες για τις πρόσφατες εξελίξεις. Ε, θα ήθελα να σας ε, τονίσω τώρα κάποια ζητήματα τα οποία δεν τονίζονται συχνά. Το πιο σημαντικό νέο για τους βουλευτές είναι ότι πριν από ένα μήνα είχαμε την κυρία Αθανασοπούλου την νέα επικεφαλής η οποία ε, μπήκε σε αυτή τη θέση πριν από ένα μήνα στην Κομισιόν και συνεργάζεται με, με την Επίτροπο Μπιενκόφσκα, είναι υπεύθυνη για αυτή την ε, μονάδα. Την έχω δει ε, τις τελευταίες εβδομάδες κάποιες φορές, ε, είναι εξαιρετική και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που ηγείται αυτής της μονάδας. Ε, κάτι άλλο σημαντικό είναι ότι το Παγκόσμιο Γραφείο Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών έκανε τη γενική του συνέλευση στην Κίνα. Όπως πάντα, εγώ εκπροσώπησα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, εξέλεξαν τον κύριο Σικασφίλη από τη Γεωργία ως πρόεδρο. Εμείς ε, ασκήσαμε πίεση εκ μέρους της, Επιστρο... της Επιτροπής ε, Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πριν από τρία χρόνια είχα προτείνει για πρώτη φορά να υπογράψουμε μία συμφωνία συνεργασίας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού Η Καρή Μαντέλη και ο κύριος ε, Ταγιάννη, η Καρή Μαντέλη και Ταγιάννη θα δεχτούν ε, τον ε, πρόεδρο στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο έχει διοργανώσει ένα πολύ σημαντικό γεγονός, μια εκδήλωση για τον τουρισμό. Εδώ έγινε. Ήταν η Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Ένα γεγονός που ενέπνευσε πολλούς Εκατοντάδες ήρθαν από παντού, από την Ευρώπη, ειδικοί οργανώσεις. Ευχαριστώ λοιπόν το επιτελείο του κυρίου Ταγιάννη γι' αυτό. Θα τα πω και αργότερα. Η Εστονική Προεδρία επίσης διοργάνωσε ένα φόρουμ εμπειρογνωμόνων για τον τουρισμό. Εκπροσώπησα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πάντοτε κάνω μια παρουσίαση βέβαια για τους στόχους και τις προτεραιότητές μας σε τέτοιες εκδηλώσεις και θα ήθελα να αναφέρω ότι στο Λονδίνο όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν εκπροσώπηση την περασμένη εβδομάδα σε μια άλλη εκδήλωση για τον τουρισμό. Είχαμε εκεί όλους τους υπουργούς ε, που είναι υπεύθυνοι για τον τουρισμό. Και θα τελειώσω με αυτό, που είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που έχουμε καταφέρει να πετύχουμε είναι το εξής. Υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί που είναι ενεργοί στον τομέα της τουριστικής ε, διπλωματίας, όπως και οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί. Τώρα εμείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πάντοτε είμαστε προσκεκλημένοι σε τέτοια διεθνή φόρα. Πραγματικά ε, αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε την φωνή μας να ακουστεί, γεγονός που δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Μπορούμε λοιπόν τώρα να, να συμμετάσχουμε σε τέτοια σε, ε, σε Υπάρχει και μια σχετική διάσκεψη για τον τουρισμό που θα λάβει η χώρα σύντομα. Αν έχετε ενδιαφέρον, μπορώ να σας δώσω τα στοιχεία. Επίση, το Νοέμβρη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διοργανώσει το γνωστό ετήσιο φόρουμ για τον τουρισμό, αν θυμάμαι καλά, είναι στις 28. Αλλά νομίζω ότι η Επίτροπος ε, θα ε, καλωσορίσει εκεί ε, οποιονδήποτε θέλει να παραβρεθεί. Όποιος ευρωβουλευτής θα είναι πρόσδεκτος. Τέλος, υπήρξαν πολλά επιτυχημένα πιλωτικά προγράμματα και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη βοήθειά σας. Έχουμε λάβει μεγάλη χρηματοδότηση. Τα project για τον τουρισμό ε, για την πολιτιστική Ευρώπη πήραν 1,1 εκατομμύριο ευρώ. Το project Interrail πήρε 12 εκατομμύρια ευρώ. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη βοήθειά σας. Τους επόμενους δύο μήνες η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα ε, πολιτισμού θα ξεκινήσει ως project και θα σας δώσω ε, στοιχεία γι' αυτό αργότερα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Ουλουρή. Ξεκινάμε αμέσως με την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, της μελέτης για τη φορολογία στον τομέα του τουρισμού. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ και που συντάξατε αυτή τη μελέτη για την Επιτροπή μας. Πρόκειται για μια ανάλυση ε, της κατάστασης της φορολογίας στον ε, τουρισμό στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάμε επίσης και κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, τις επιπτώσεις στην οικονομία. Δίνω το λόγο στον καθηγητή, ο οποίος ε, θα μας παρουσιάσει την έκθεση. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Έχετε το λόγο για 8 με 10 λεπτά ακριβώς. Θα βάλω χρονόμετρο, γιατί έχουμε καθυστερήσει λίγο. Είμαι βέβαιη όμως ότι θα κάνετε μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα δούμε μόνο τα βασικά των εργασιών μας επειδή μας πιέζει ο χρόνος. Λέγομαι Σάιμον Κέρι Είμαι από την Price Waterhouse Keepers και είμαι ε, σύμβουλος πολιτικής. Ήμουν πρώην σύμβουλος ε, του Υπουργείου Οικονομικών ε, και εγώ είμαι ο Τζόναθαν Κίλαμ, οικονομολόγος στο οικονομικό τμήμα της Price Waterhouse. το μερίδιο του τουρισμού το οποίο ε, αναλογεί στην ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση σε παγκόσμιο επίπεδο έχει πέσει ουσιαστικά, έχει μειωθεί σημαντικά. Σταθεροποιήθηκε τα τελευταία πέντε χρόνια περίπου στο 40% του παγκόσμιου τουρισμού αλλά 20 με 30 χρόνια πριν ήταν σχεδόν στο 55% το ποσοστό ο αριθμός των τουριστών που επισκέπτονται την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυξανόμενος. Δεν υπάρχει μία εξήγηση για τη μείωση στο μερίδιο του παγκόσμιου τουρισμού. Η αγορά του παγκόσμιου τουρισμού αυξάνεται και οι άνθρωποι ε, όσο πλουτίζουν πηγαίνουν και σε μεγαλύτερες ε, αποστάσεις ε, και σε νέους προορισμούς και αναδύονται και νέοι προορισμοί συνεχώς. Υπάρχει όμως και το γεγονός ότι το ισοζύγιο του τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σταθεροποιηθεί τα τελευταία πέντε χρόνια και ένας λόγος γι' αυτό είναι ε, κάποια θέματα ασφαλείας στις γειτονικές χώρες. Για παράδειγμα, άνθρωποι που θα πήγαιναν στην Τουρκία ή σε κάποιες χώρες της Βόρειας Αφρικής. Τώρα πλέον δεν κάνουν αυτά τα ταξίδια και ε, ταξιδεύουν ε, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταυτών. Το ευρωπαϊκό λοιπόν μερίδιο του παγκόσμιου τουρισμού έχει μειωθεί μεν, αλλά σταθεροποιήθηκε, αλλά ο αριθμός των τουριστών που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνονται. Πολύ σύντομα, η μελέτη που έγινε ε, κατόπιν παραγγελία τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέτασε τέσσερα στοιχεία. Έδωσε μια βάση δεδομένων ε, για τον ε, τομέα του τουρισμού στα κράτη-μέλη. Εξετάσαμε κάποιες περιοχές ως δειγματοληπτικές μελέτες, έγινε ανάλυση και κάναμε και κάποιες γενικές συστάσεις ε, για την φορολόγηση του τουρισμού εν γέννη. Ε, κυρίως κοιτάμε να δούμε τι είδου φορολόγηση θα έχουμε, ε, φόρο διαμονής ή φόρο με τη μορφή του ΦΠΑ για παράδειγμα. Δεν θα επισέλθω σε πάρα πολλέ ε, λεπτομέρειες για τη βάση δεδομένων, θα δημοσιευτεί, θα τη δείτε κάποια στιγμή. Δεν μας εξέπλεψε βεβαίω το γεγονός ότι υπάρχει ε, μεγάλη διαφοροποίηση στον τρόπο φορολόγηση. Υπάρχουν ε, προσωπική φορολόγηση, ΦΠΑ, τέτοιες μορφής φόροι και αν δούμε συγκεκριμένα φόρο διαμονής Αυτά αφορούν ε, διαμονή βραχίας διάρκειας ε, σε ξενοδοχεία για παράδειγμα και εφαρμόζονται παγκοσμίω. Αρχικά ήταν αμερικανικό φαινόμενο, τώρα υπάρχουν παντού τα δύο τρίτα των κρατών μελών αυτή τη στιγμή ε, εφαρμόζουν τέτοιο φόρο διαμονής και ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται αλλάζει ε, ανάλογα με τη χώρα. Ορισμένες φορές ε, είναι ένας φόρος ο οποίος δίνεται φάπαξ, ορισμένες φορές εφαρμόζεται μέσα στην τιμή κλπ. Θα ήθελα να σταθώ στο ΦΠΑ γιατί είναι πολύ σημαντικός φόρος για τον κλάδο και όπως γνωρίζετε τα περισσότερα κράτη-μέλη ούτως ή άλλως εφαρμόζουν μειωμένο ποσοστό ΦΠΑ για τις τουριστικές υπηρεσίες, ε, διαμονή, ε, μεταφορές κλπ. Τα κράτη-μέλη έχουν μικρό περιθώριο να μειώσουν περαιτέρω το ΦΠΑ. Αν ε, δείτε για παράδειγμα το ΦΠΑ στη διαμονή, τα μισά κράτη-μέλη ήδη ούτως ή άλλως έχουν το μικρότερο ποσοστό σε αυτή την περίπτωση, επομένως πόσο πιο κάτω να πάει. Μετά τη βάση δεδομένων λοιπόν, με βάση τα στοιχεία που είχαμε, είδαμε τα φορολογικά συστήματα τριών πολύ επιτυχημένων τουριστικών ε, προορισμών. Είδαμε την Κύπρο συνολικά ως χώρα. Η Κύπρος είναι ενδιαφέρουσα γιατί εφαρμόζει πολύ χαμηλή φορολογία ε, γενικά στην οικονομία της αλλά κυρίως και στον τομέα του τουρισμού και η κυβέρνηση κάνει διαφοροποίηση στις προσφορές ε, και στη φορολόγηση του τουρισμού. και έχουμε τουρισμό ε, πολύ εξειδικευμένο σε κάποιες περιπτώσεις, ε, τουρισμό πολυτελείας κλπ. Είδαμε επίσης ε, τι τις νήσου, νήσους, τη Μαγιόρκα, τη Μενόρκα και την Ήμπιζα, όπως και την Κύπρο έχουν πολύ χαμηλή ε, φορολόγηση και είναι της, ε, περιφερεια... της αυτόνομης περιφέρειας οι φόροι και πρόσφατα έχουν και ένα νέο το φόρο διαμονής και βιώσιμου τουρισμού που είναι αντίστοιχο με ένα φόρο ο οποίος εισήχθη πριν από 15 χρόνια και ανακλήθηκε ένα χρόνο αργότερα για διάφορου λόγου και εξετάσαμε τι διαφορά είχαν οι δύο αυτοί φόροι και υπάρχουν ε, αρκετά στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν ότι ο τρόπος με τον οποίο εισήχθησαν και στη συνέχεια έγινε διαχείριση αυτών των φόρων ήταν τελείως διαφορετικός και υπήρχε και αντίστοιχη υποδοχή. Και τέλος εξετάσαμε το Παρίσι ως πόλη, πολύ δημοφιλής προορισμός. Το Παρίσι εφαρμόζει διάφορους φόρους στον τουριστικό τομέα και για το Παρίσι ιδιαίτερα ο τομέας της ε, διαμονής είναι πάρα πολύ σημαντικός, ε, Airbnb, το Away και άλλες πλατφόρμες που παρέχουν ε, υπηρεσίες έχουν πολύ μεγάλη παρουσία εκεί. Το Παρίσι ήταν ε, από τις χώρες που εφέρμοσαν ε, πολύ γρήγορα το μοντέλο στο οποίο εφαρμόζεται ο φόρος από τον πάροχο της πλατφόρμας και όχι από τον ίδιο τον ξενοδόχο ή τον ιδιοκτήτη του κύματος στο οποίο παρέχει διαμονή και να δώσω τώρα το λόγο στον συνάδελφο. Θα σας πω κάποια βασικά απορίσματα σε οικονομικό επίπεδο που έχουμε από τη μελέτη. Ε, το οικονομικό αποτύπωμα που αφήνει ο τομέας του τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ουσιαστικό. Είναι χονδρικά το 5% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ και αν ε, προσμετρήσουμε εδώ και τις ε, βασικές σχέσεις της αλυσίδας προμηθειών του τουρισμού πηγαίνουμε περίπου στο 10%. Για χώρες όπως η Ελλάδα, ο τομέας του τουρισμού είναι το 18% χονδρικά του ΑΕΠ της χώρας, είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικός τομέας. Αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία ε, για το για ποιο λόγο παραμένει κάποιο εντό Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καταρχά ε, οι τιμέ, αλλά δεν είναι μόνο οι τιμέ των ξενοδοχείων, αλλά και άλλα σχετικά. Ε, ε, σχετικέ υπηρεσίε, ενοικιάσει αυτοκινήτων, ε, τιμέ στα εστιατόρια κλπ. Αλλά και η ποιότητα. Όταν αναφερόμαστε στην ποιότητα, ε, κυρίω αυτό αφορά κοινωνική ανάπτυξη, σχετικέ υποδομέ και ποιότητα του περιβάλλοντο. Και αυτά συμβάλλουν ώστε να υπάρχουν μοναδικοί προορισμοί, του οποίου θέλει να επισκεφθεί ο τουρίστα. Οι φόροι διαμονής είναι πολύ χαμηλοί, είναι ε, από, ένα, ε, από 50 cent μέχρι 7,5 ευρώ τη βραδιά ε, στις πολύ υψηλέ χρεώσεις αλλά δεν είναι τόσο υψηλή ώστε να αποτελούν ένα σταλτικό παράγοντα και να μην θέλει ο τουρίστας να παραμείνει όταν προσφέρονται δε πολύ δελεαστικά πακέτα. Σε προορισμούς βέβαια που υπάρχει μικρότερη ζήτηση που δεν υπάρχουν κάποια καλά στοιχεία ποιότητας θα δείτε πολύ πιο σημαντικές συνέπειες τέτοιων φόρων διαμόρφωσης ή τουρισμού εν Όσον αφορά τις συστάσεις της έκθεσής μας, αυτό το οποίο θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι όταν οι τουρίστες ε, έρχονται εκτό Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικό και για το συνάλλαγμα ε, στις ε, οικονομίες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28. Η φορολόγηση είναι παράγωνο ο οποίος γεννά συνάλλαγμα αλλά θεωρείται ότι στρεβλώνει την αγορά και η μείωση των τιμών προσθέτουν πάρα πολλά στην ευρωπαϊκή οικονομία, κυρίως για να αποτελεί ε, ελκυστικό προορισμό. Και επίσης, οι προορισμοί που μπορούν να υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαφέρουν από διάφορους άλλους παγκόσμιους τορισμούς. Ε, όσο πιο ισχυρή γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προορισμός θα μπορέσει να ανατρέψει και κάποιες από τις ε, τάσεις μείωσης που είχαμε. Να πω δύο λόγια τώρα όσον αφορά τον ε, φόρο διαμονής, ε, τον BETAX. Ε, διαφέρει ο τρόπος που εισάγονται και γίνεται η διαχείρισή τους. Για παράδειγμα, αν δείτε τις Βαλεαρίδες νήσους, ε, ο τομέας συμμετείχε στη διαδικασία διαβούλευσης καταλήλως τα έσοδα ε, κρατούνται για τον κλάδο και αυτό φυσικά ε, δημιουργεί και περαιτέρω διαφάνεια και ο κλάδος συμμετέχει και στις τελικές αποφάσεις. Ε, υπάρχει δηλαδή πολύ μεγάλη συνένεση για την εφαρμογή του συγκεκριμένου φόρου οι φόροι αυτοί διαμονής σε γενικέ γραμμές είναι ε, ευθύνη των ε, ξενοδόχων ή αυτών που παρέχουν τη διαμονή ε, και αυτοί θα πρέπει να του συλλέγουν και από εκεί πέρα να αποδίδονται αλλά υπάρχουν και κάποια θέματα συμμόρφωσης. Ουσιαστικά ζητάτε από τους ξενοδόχους να είναι φοροεισπράκτορες και αυτό ε, αρχίζει βέβαια και βελτιώνεται σε περιοχές για παράδειγμα όπου στο Παρίσι ο πάροχος ε, της πλατφόρμας είναι αυτός ο οποίος συλλέγει το φόρο. Ε, δεν θα πω πολλά για τις συστάσεις γιατί μας τελείωσε ο χρόνος, αλλά η έκθεση είναι διαθέσιμη και σας προτρέπω λοιπόν να δείτε τα συμπεράσματά μας και τις συστάσεις μας ιδιαίτερως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Θα ξεκινήσει η συζήτηση τώρα. Ο κύριος Ντεγκράντες Πασκουάλ. Έχετε το λόγο. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για την παρουσίαση αυτή, παρά το γεγονός ότι ήταν γενική παρουσίαση. Θα ήθελα να πω όμω κάτι το οποίο έχω επαναλάβει αρκετέ φορέ εδώ στην Επιτροπή. Ευτυχώ ε, ήταν ε, έξυπνη συνθήκη και δεν απέτρεψε την εναρμόνιση σε θέματα τέτοια ε, φορολογίας τουρισμού. Ό,τι αφορά λοιπόν τη φορολογία δίνει και ένα ε, περιθώριο ελευθερίας και αυτό επιτρέπει την ανταγωνιστικότητα ε, σε ένα κλάδο όπως είναι ο τουρισμός ε, που είναι πάρα πολύ σημαντικός για κάποιες χώρες. Σίγουρα για τη δική μου, για την Ισπανία, ο τουριστικός κλάδος είναι ο πρώτος στη χώρα και Αντί να μειώνονται οι ε, ποσοστώσεις, αυξάνονται καθημερινά. Η φορολογία του τουρισμού ε, έχει ε, σημασία ε, κυρίως για μια χώρα που είναι τουριστικός προορισμός. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι φόροι είναι τελείως διαφορετικοί από τους δασμού. δεν είναι ακριβώς το ίδιο ε, σε επίσημο, ε, σε τυπικό επίπεδο και συνήθως ε, οι φόροι αυτοί που χρησιμοποιούνται και κυρίως είναι απαραίτητη για τον τομέα της παροχής τουριστικών υπηρεσιών. Εγώ είμαι κατά ε, των φόρων για τις τουριστικές υπηρεσίες που ξεκίνησαν από τις Ηνωμένε Πολιτείε που μετά όμως μετατράπηκαν σε ιδεολογικό φαινόμενο πολλές φορές με την αιτιολογία ότι με αυτούς τους φόρους ε, ε, πληρώνονται περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργούνται από τον τουρισμό. Αυτό δεν ισχύει. Και μάλιστα κάποιος μας ενημέρωσε ότι στις Βαλεαρίδες Νήθους είχαμε το εξή, μας είπατε ότι στην αρχή εισήχθη ο φόρος, μετά ε, αποσύρθηκε και μετά επανεισήλθε. Είναι καθαρά ιδεολογικό το θέμα. Ε, τον επέβαλε μια κυβέρνηση αριστεράς, ε, την απέσυρε η κυβέρνηση του ΕΛΚ και τώρα του Λαϊκού Κόμματος, και μετά τον επανεσήγαγε και πάλι μια αριστερή κυβέρνηση. Νομίζω λοιπόν ότι είναι για ιδεολογικούς λόγους αυτή η φόρη. Τον εφαρμόζουμε φόρους για ε, τουριστικές υπηρεσίες ε, για μένα είναι λανθασμένο. Μια χώρα που χρησιμοποιεί τον τουρισμό για να αυξήσει το ΑΕΠ της και να αυξήσει και την απασχόληση και τον πλούτο της... Ε, πέραν των θετικών κινήτρων που πρέπει να έχει για τον τουρισμό, θα πρέπει να προσπαθήσει ε, για να μην ε, δημιουργήσει και ε, προβλήματα και να μην είναι ανασταλτικός παράγων η εφαρμογή του τουρισμού. Γιατί πολλές φορές ο πελάτη αναρωτιέται γιατί του επιβάλλει το ξενοδοχείο φόρο διαμονής. Αλλά δεν είναι το ξενοδοχείο αυτό που τον επιβάλλει. Τον επιβάλλουν ε, οι κυβερνητικέ αρχέ. Ευχαριστούμε. Πολύ λίγο χρόνο μου δώσετε. Δεν μπόρεσα να εκφράσω τι απόψει μου. Ναι, αλλά έχουμε καθυστερήσει. Και πρέπει κι άλλοι να πάρουν το λόγο. Η κυρία Μπιλμπάου. Ναι, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και θα ήθελα να ε, ε, συγχαρώ τον Μπιλμπάου γιατί εχθές ε, έλαβε το βραβείο τη καλύτερη πόλη του 2018. Σας καλούμε λοιπόν όλους να επισκεφτείτε την πόλη του Μπιλμπάου που πλέον έχει και αυτό το βραβείο και σίγουρα θα περάσετε πολύ καλά. Να σας ευχαριστήσω για την έκθεσή σα. Για μας ε, το φαινόμενο του τουρισμού στη χώρα των Βάσκων ε, είναι νέο φαινόμενο. Μας ανακαλύπτουν νομίζω σιγά σιγά εδώ τα τελευταία χρόνια και όλο ο κόσμο γνωρίζει το γιατί, γιατί έχουμε μια πρόσφατη ιστερία πολύ σκληρή και ζωφερή και χαιρόμαστε που επιτέλους μας βλέπουν με άλλο μάτι. Ε, όσον αφορά τους φόρους και τους δασμούς που επιβάλλονται, Πρόκειται για μια συζήτηση η οποία είναι ακόμα ανοιχτή και αυτό το οποίο θα μπορούσα να σας πω είναι ότι στους ε, χώρους ε, που βλέπουμε ότι ε, εμφανίζεται ένα φαινόμενο το οποίο δεν γνωρίζαμε, ε, αρχίζουμε να σκεφτόμαστε πάρα πολύ τι είδους φόρους και δασμούς θα μπορούσαμε να επιβάλλουμε, όχι τόσο για να μειώσουμε το φαινόμενο και να μειωθούν οι τουρίστες που θα μπορούσαν να έρθουν στις περιοχές μας, αλλά κυρίως εν μέρη και γιατί θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να διατηρήσουμε την ποιότητα, αυτή το βιώσιμο τουρισμού που νομίζω ότι αυτό είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να επιδιώκουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, δεν έχει τόσο σημασία αν θα είναι υψηλό ή χαμηλό ο φόρο. Θα πρέπει να προσπαθούμε να έχουμε βιωσιμότητα και τουρισμό ποιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί είδαμε και τι συνέπειε σε κάποιε περιοχέ τι οποίε δεν έγινε σωστή δουλειά. Μαζικό τουρισμό, ο οποίο δημιουργεί ζημίε, δημιουργεί προβλήματα και δεν είναι τα πάντα οικονομία στο ευρωπαϊκό μοντέλο. Όπως και να έχει, αυτό το οποίο σίγουρα θα ήθελα να πω και δεν είχα χρόνο να δω και τι συστάσεις είναι ότι εάν ε, επιβάλλεται στα ξενοδοχεία να συλλέγονται αυτός ο φόρος, ε, σίγουρα ο φόρος αυτός θα πρέπει να είναι ένας φόρος ο οποίος ε, θα πρέπει να έχει και ένα χαρακτήρα για κάποιο σκοπό. Δηλαδή δεν το βλέπουμε. Συλλέγεται αυτός ο φόρος από ένα ξενοδοχείο και μετά τι γίνεται με αυτό το φόρο. Σίγουρα δεν είναι όλες οι περιοχές ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάποιες, κάποιοι θα επιλέξουν να κάνουν καλύτερα πράγματα για την περιοχή ώστε να είναι πιο δελαστικός ο προορισμός. Κάποιοι άλλοι έχουν να διορθώσουν πράγματα. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιοι ελάχιστοι κανόνες εναρμόνισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ουσιαστικό είναι να συλλέγονται οι φόροι για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό για τον τουρισμό. Να βοηθούν τον τουρισμό. Η κυρία Αρνούτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε βλέπω στην μελέτη την σχέση που υπάρχει μεταξύ χαμηλής φορολογίας και της προσέλκυσης των ε, τουριστών. Αυτό είναι κάτι που δεν είναι καινούριο βεβαίως. Έχω μία ερώτηση. Πόσο στήχησε αυτή η μελέτη της ε, Price Waterhouse Cooper στον Ευρωπαίο καταναλωτή. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Ποια είναι η σκοπιμότητα. Όλα πρέπει να τα κάνουμε ομοιόμορφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται όμως για αρμοδιότητα των κρατών μελών και των δικών τους διοικητικών αρχών. Από την άλλη, οι πλατφόρμες τύπου Uber και Airbnb κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μην ε, υποβληθούν σε οποιαδήποτε φορολογία και αν το καταφέρουμε να τους φορολογήσουμε αυτό είναι πραγματικά εξαίρεση. Αυτό λοιπόν που μας ενδιαφέρει εδώ είναι πρώτον να δούμε κατά πόσον οι αποφάσεις αυτές μπορούν να εφαρμοστούν σε εθνικό επίπεδο και μετά να κοιτάξουμε τις αποφάσεις αυτές επί της ουσίας. Το βασικό πρόβλημα σήμερα στον τουρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το θέμα της ασφάλειας. Στη Γαλλία αυτό το είδαμε. Δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τους ε, τουρίστες οι οποίοι θέλουν να επισκεφτούν τη χώρα μας και ίσως θα ήταν λίγο πιο ενδιαφέρον όχι μόνο να γίνει μελέτη αλλά να διαπιστώσουμε ότι και εδώ πρόκειται για αρμοδιότητες εθνικές και αρμόδια για την ασφάλεια των τουριστών είναι ακόμα τα κράτη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Εύενς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ πραγματικά χαιρετίζω αυτή την έκθεση που εκπροσωπεί εδώ πολλές περιοχές όπως την Ουαλία. Είμαστε σήμερα σε μια νέα κατάσταση όσον αφορά την τοπική φορολογία και μάλιστα σε περίοδο διαβούλευσης καλούνται οι πολίτες της περιοχής μας να αποφανθούν όσον αφορά την μορφή της φορολογίας και το ύψος. Βεβαίως πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο θέμα. Υπάρχει αντιπολίτευση, υπάρχει αντίσταση και η μείωση του ΦΠΑ παραδείγματος χάρη είναι κάτι που σαφώς ε, ενδιαφέρει τον τουριστικό τομέα στην Ουαλία αλλά και σε άλλες περιοχές, στη Σκοτία και αλλού που δεν υπάρχουν τέτοιου είδους φόροι όπως ε, αυτοί που ισχύουν σε άλλες περιοχές για τις ε, διαμονές, για τα ξενοδοχεία. Όπως διαβάζουμε και στην έκθεση, υπάρχουν κάποιες ε, περιοχές που σίγουρα όπως η Ουαλία μπορούν να επιβάλλουν έναν μικρό φόρο χωρίς αυτό να έχει άμεσες επιπτώσεις στις κρατήσεις και στον αριθμό των τουριστών. Βεβαίως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί είδαμε και περιπτώσεις όπου οι τουρίστες τράφηκαν σε άλλες περιοχές, εκεί δηλαδή που δεν υπήρχε καμία φορολογία. Είναι πολύ σημαντικό επίσης η Task Force η οποία επεξεργάζεται το θέμα αυτό να κοιτάξει πώς ακριβώς μπορούν να κατανεμηθούν τα ε, ποσά αν υπάρχει παραδείγματο χάρη αρκετή έμφαση που δίνεται στην βιωσιμότητα, στον αηφόρο τουρισμό, γιατί αυτά είναι θέματα τα οποία δεν βρίσκονται στο πρώτο επίπεδο του ενδιαφέροντος έκθεση αυτή. Βεβαίως και τίθενται σωστά ερωτήματα, αλλά ίσως δεν έχει πάει ακόμα αρκετά βαθιά αυτή η έκθεση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Εύαν, λέει η Πρόεδρος, οι εμπειρογνώμονε. Μπορείτε να δώσετε κάποιες απαντήσεις. Και έχω και μια άλλη ερώτηση εγώ. Πώς υπολογίζετε τη φορολογία Από ό,τι κατάλαβα, λέτε, βασίζουμε το φόρο στον αριθμό των ε, δωματίων. Όσον αφορά όμως τη φορολόγηση Airbnb, εκεί ποιο είναι η μονάδα μέτρησης. Είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστεί εκεί η φορολογία. Ποια είναι η μέθοδό σας και ποιες είναι οι παράτημοι. Δυστυχώς έχετε μόνο δύο λεπτά. Γιατί έχουμε και μια άλλη μελέτη που πρέπει να επεξεργαστούμε. Έχετε το λόγο. Ναι. Ο φόρος αυτός διαμονής γίνεται όταν γίνει η κράτηση και η πλατφόρμα ουσιαστικά υπολογίζει τον ε, φόρο και τον ε, συνυπολογίζει στην τιμή που πληρώνει ο τουρίστας που κάνει την κράτηση. Στα ξενοδοχεία γίνεται μια διαφορετική τιμολόγηση και υπάρχει μια ξεχωριστή, ε, θα έλεγα, καταγραφή του φόρου διαμονής. Ο τουρίστας την ώρα που πληρώνει το δωμάτιό του και φεύγει από το ξενοδοχείο, πληρώνει το φόρο διαμονής ξεχωριστά, εάν έχει προπληρώσει την κράτηση. Τώρα, εάν αυτός ο φόρος διαμονής είναι ή δεν είναι μειονέκτημα και μπορεί να οδηγήσει κάποιους τουρίστες από το να στραφούν σε άλλες περιοχές που δεν επιβάλλεται η φορολογία. Όπως ακούσατε, αυτή η φόρη είναι σχετικά χαμηλή, είναι τουλάχιστον χαμηλή σε σχέση με την συνολική τιμή που πληρώνει ο τουρίστας και βεβαίως βλέπουμε ότι η κατανομή αυτού του φόρου στις διάφορες περιοχές ε, γίνεται με εμαλό τρόπο. Στην ε, Μεσόγειο, στην ε, Νότια Ευρώπη, εκεί που υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, σίγουρα μπορεί να υπάρχει μια επίπτωση της φορολογίας. Εγώ θέλω να υπογραμμίσω δύο σημεία. Πρώτον, το πόσο μοναδικές είναι οι περιοχές και για ποιο λόγο ο τουρίστας επιλέγει να πάει σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό δίνει τη δύναμη σε κάποιους συγκεκριμένους τουριστικούς προορισμούς να επιβάλλουν μια φορολογία. Βεβαίως ε, χρειάζεται προσοχή έτσι ώστε η φορολογία αυτή να είναι διαφανής και να είναι σαφές πότε επιβάλλονται και ποιο ακριβώς είναι το ύψος τους. Τέλος, για να προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιες από τις παρατηρήσεις που έγιναν, η φύση αυτής της φορολογίας είναι χαμηλή. Οι οικονομικές επιπτώσεις της είναι πολύ ε, μηδαμινές. Γι' αυτό και επαναλαμβάνουμε ότι πρέπει να καταλάβετε ότι όταν επιλέγει ένας τουρίστας μεταξύ πολλών προορισμών, εκεί μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο η φορολογία, αλλά για αποφασισμένους τουρίστες, τουρίστες οι οποίοι θέλουν να πάνε σε ένα μοναδικό μέρος, εκεί πραγματικά ο παράγοντας φόρος διαμονής δεν είναι τόσο σημαντικός. Όσον αφορά την αρμοδιότητα ε, των κρατών μελών, ναι, συνεχίζει να είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ολοκληρώσαμε την επεξεργασία της πρώτης μελέτης. Νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στην δεύτερη, που αφορά τον ναυτικό τουρισμό. Ο κύριος Λέμαν θα μας παρουσιάσει το έγγραφο καλωσορίσατε παρουσιάζει τις ε, δυνατότητες και τις δυσκολίες του ναυτικού τουρισμού στον ε, τομέα αυτό. Θα μιλήσουμε για τις άδειες, για τα λιμάνια, για τον εξοπλισμό ασφάλειας, για την κυκλική οικονομία και βεβαίως για τη νέα τεχνολογία που εφαρμόζεται στον τομέα αυτό. Κύριε Λέμαν, είστε επικεφαλής της ε, μπλε οικονομίας του θαλάσσιου σχεδιασμού και έχετε ακριβώς 7 λεπτά. Έχετε το λόγο. Bien sûr, ça va, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα αγγλικά. Εκτός μικροφώνου του σχολείου της Πρόεδρου. Ξέρω, αλλά έχω ετοιμαστεί, προετοιμαστεί στα αγγλικά και είναι και πιο εύκολο να μιλήσεις 7 λεπτά στα αγγλικά. Ο παράκτιος ε, και ναυτικός τουρισμός, ε, παραθαλάσσιος τουρισμός, είναι ένας από τους βασικούς ε, τομείς που έχουν επιλογή από την πλέον στρατηγική της Κομισιόν για το 2012. Το 2014 υπήρξε η στρατηγική γενικά για τον ε, παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό η οποία είχε στόχο να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και την βιωσιμότητα του τομέα, την δημιουργία θέσεων εργασίας, γενικά ό,τι ε, επιδιώκουν και όλες οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κομισιόν. Έχουμε λοιπόν τέσσερις πυλώνες, ε, ανταγωνιστικότητα, δεξιότητες, καινοτομία, βιωσιμότητα και φυσικά μεγιστοποίηση της χρηματοδότησης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας δούμε τώρα κάποιους υποτομείς ε, του να ξεκινήσω λέγοντας βέβαια ότι αυτός ο τομέας είναι ένας από τους μεγαλύτερους ε, στην Ευρώπη. Είναι το 1 τρίτο της ε, ναυτικής οικονομίας, της θαλάσσιας ε, οικονομίας, 23 δις ευρώ σε προστιθέμενη αξία. Αν δείτε τον υποτομέα του ναυτικού τουρισμού τώρα, ένας τους 10 πολίτες ε, κάνει θαλάσσια σπορ τακτικά, κανό, ιστιοπλοεία, σέρφινγκ, ε, καταδύσεις, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. 36, 36 ε, εκατομμύρια πολίτες έχουν σκάφη και έχουμε πολλά εκατομμύρια σκάφη στα ευρωπαϊκά ύδατα. Έτσι λοιπόν ο τζίρος είναι 6 δις ευρώ. Έχουμε 20.000 θέσεις εργασίας ε, στον τομέα των ε, ναυλώσεων και οι ευρωπαϊκές μαρίνες έχουν 4 ε, δις ευρώ σε τζίρο και απασχολούν μεταξύ των 40 και 70.000 ανθρώπων. Είναι δύσκολο να το πει κανεί ακριβώς αυτό το νούμερο, γιατί είναι μικροεπιχειρήσεις οι μαρίνες και είναι δύσκολο κανείς να μετρήσει πόσοι απασχολούνται εκεί. Ο τομέας όμως έχει και κάποιες προκλήσεις να αντιμετωπίσει έχουμε δει μια αύξηση ε, της ηλικίας των σκύπερα από τα 45 στα 54 έτη μέσα στα τελευταία περίπου 10 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι πολλοί νέοι οι οποίοι μπήκαν στο χώρο για προφανείς λόγους. Η 30 ε, χρόνια είναι η ζωή των ε, σκαφών, των γιότ, με πλαστικά ενισχυμένα και ε, fiberglass, όλα αυτά τώρα έχουν αλλάξει ε, βέβαια την τεχνολογία, αλλά όπως και να έχει είναι γυρασμένος ο στόλος και θα έρθω σύντομα στις λύσεις. Επίσης υπάρχουν διάφορα ενδιαφέροντα ε, ανάμεσα στους τουρίστες. Θέλουν να έχουν συνεχώς κάτι διαφορετικό, να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τους συσκευές, όπως είδαμε και με το CITS και τις μεταφορές. Άρα αυτό το έγγραφο έχει επικεντρωθεί στα τέσσερα στοιχεία που μόλις ανέφερε και η Πρόεδρος. Μιλάμε για τις ε, άδειες, ε, για τους ε, για τον εξοπλισμό, για την ανακύκλωση των σκαφών κτλ. Ε, κάτι που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι πλέον ο κόσμος δεν αγοράζει σκάφη, αλλά μισθώνει, ναυλώνει. Οι επαγγελματίες skippers, ε, αδειοδοτημένοι skippers, δεν αναγνωρίζονται αυτόματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό σημαίνει απώλεια εισοδήματος. Αν θέλει κανείς να αναβλώσει μια εταιρεία για παράδειγμα να αναβλώσει και να ε, αποσχολήσει κάποιον για την ε, υψηλή περίοδο δύσκολα βρίσκει ανθρώπους. Ε, υπάρχει ένα project για τη σύγκριση των αδειών κοιτώντας τα βασικά τους προσόντα, όμως σε αυτή τη μελέτη ακόμα έχουμε συμπεριλάβει μόνο μερικά κράτη-μέλη. Ευχαριστούμε τον κύριο Νταγκιγιάρ που στην ουσία έχει πιλωτάρει αυτό το project που θα ξεκινήσουμε για τους skippers. Επόμενη διαφάνεια. Δείχνει ακριβώς δύο πανομοιότητα σκάφη με δύο διαφορετικές σημαίες. Ο skipper μπορεί να οδηγήσει μόνο ένα από τα δύο, ακόμα και αν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Μετά, κοιτάξαμε ένα άλλο πρόβλημα για τον εξοπλισμό που έχει να κάνει με την ασφάλεια των σκαφών. Είναι θέμα εσωτερικής αγοράς. Έχουμε τους εθνικούς κανόνες, τους ευρωπαϊκούς κανόνες και τον, τους κανόνες των ε, κρατών στα οποία θα πλεύσουν τα σκάφη. Άρα έχουμε την ίδια συσκευή αλλά διαφορετική εκτέλεση της νομοθεσίας γιατί στην ουσία δεν συμμορφώνεται η συσκευή με την νομοθεσία ε, σε όλα τα κράτη. Ε, αυτό που ζητάμε λοιπόν είναι είτε να τηρούνται μόνο οι απαιτήσει του κράτου σημαία και τα άλλα κράτη να μην ζητούν εφαρμογή, αλλά ε, φυσικά να υπάρχουν κάποια minimum standards στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε και μια τυποποίηση των κανόνων. Το τρίτο στοιχείο είναι η ανάπτυξη των μαρινών και της χρήσης των σκαφών. Συνήθως οι μαρίνες χρησιμοποιούνται για αποθήκευση των σκαφών. όπω και πολλέ φορέ ε, αφήνουμε τα αυτοκίνητα στου δρόμου, εκεί να στέκονται, έτσι κάνουμε και με τι μαρίνε και τα σκάφη. Είναι μικρέ επιχειρήσει και είναι δύσκολο να του συγκεντρώσουμε. Ε, ε, σκεφτήκαμε να φτιάξουμε ένα φόρμ για να κάνουμε πιο έξυπνες τις μαρίνες και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές, αλλά είναι δύσκολο να γίνει. Οι μαρίνες έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν. Η ψηφιοποίηση θα τις κάνει πιο έξυπνε, θα γίνουν κέντρα ε, άντλησης κέρδους ε, για την ενδοχώρα και θα είναι και σύνδεσμος για άλλα προϊόντα. Ας πούμε, στο παρελθόν είχαμε μία, ε, δύο διαγωνισμούς για ναυτικούς δρόμους. Ένας που έχει να κάνει με την πολιτιστική κληρονομιά και ένας για την συνοριακούς ναυτικούς δρόμους. Το τελευταίο θέμα έχει να κάνει με την ανακύκλωση των σκαφών. 80.000 σκάφη φτάνουν στο τέλος της ζωής τους ε, ε, κάθε χρόνο. Μόνο τα 2.000 παροπλίζονται, ενώ τα υπόλοιπα μένουν έτσι στις ακτές, ε, στο νερό και ψαπίζουν. Θα, υπάρξει κάποιο, θα υπάρχει κάποιος λόγος και κάποιος τρόπος να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα παλιά σκάφη. Πρέπει όμως σε ευρωπαϊκό επίπεδο να συντονιστούμε για να τα συγκεντρώσουμε. Γιατί αυτό θα συμβάλλει και στην κυκλική οικονομία. Ε, η μελέτη έχει και κάποια συμπεράσματα, αλλά στην ουσία επαναλαμβάνουν αυτά που μόλις είπα, οπότε θα σταματήσω εδώ. Merci. Ευχαριστώ πολύ. Θα ανοίξω τώρα τη συζήτηση. Σημειώνω. Mm. Mm, mm, Monsieur De Κύριε De να είστε σύντομος αυτή τη φορά γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ και να ευχαριστήσω και τους συντάκτες της έκθεσης, ε, την οποία θα πρέπει να διαβάσουμε διεξοδικότητα, διότι περιλαμβάνει πολλά και σημαντικά στοιχεία Όλοι γνωρίζουμε ότι ο ε, παράκτιος ε, και ναυτικός τουρισμός αποτελεί πολύ σημαντική πτυχή εσόδων ε, και απασχόλησης για τις χώρες που διαθέτουν τον τουρισμό, αλλά όπως έλεγε η κυρία Μπιλμπάου για παράδειγμα, η πόλη του Μπιλμπάου που δεν έχει ακτή ε, και ε, κλίμα ε, μεσογειακό έγινε πολύ σημαντικός προορισμός τουρισμού για την κουζίνα της, για την ιδιαιτερότητά τους. Επομένως μπορεί να γίνουν και σε διάφορους άλλους, για διάφορους άλλους λόγους σημαντικός τουρισμός. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια φαινόμενα που έχουμε στον τουρισμό του ήλιου και της παραλίας που θα μπορούσε να είναι και πολύ σημαντικά υπάρχει ε, η φήμη του σεξ και του αλκοόλ οι πολλές φορές εισβάλλουν εγώ δεν είμαι κατά ούτε του σεξ ούτε του αλκοόλ σας το λέω αυτό αλλά αυτό το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι δημιουργείται στρέβλωση υπάρχουν βανδαλισμοί και ορισμένες φορές οι πόλεις ε, βιώνουν πολύ συχνά αυτοκτονίες πολύ δύσκολες ε, καταστάσεις είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Τώρα, υπάρχουν επίσης και κάποιες ε, ε, παράνομες διαδικασίες, παρατυπίες, ε, εκμεταλλεύονται κάποιοι ε, τα νέα φαινόμενα ε, του τουρισμού χαμηλού κόστους και δημιουργείται και λαφραίος τουρισμός σε διαμερίσματα και δημιουργεί και αθέμητο ανταγωνισμό σε σχέση με τα ξενοδοχεία και τις υπηρεσίες που παρέχονται οι οποίες γίνονται με καταβολή φορολογίας. Υπάρχουν επίσης και κάποιοι οποίοι απορρίπτουν τον τουρισμό. Οι μεγάλες πόλεις λένε ότι ε, πρέπει να δει κάποιο στη Ρώμη τρει ταξιμερώματα γιατί είναι αδύνατο να κυκλοφορήσει άλλη ώρα. Δημιουργούνται δηλαδή αδύνατε συνθήκε ορισμένε φορέ και αυτό αποτελεί πολύ μεγάλη συζήτηση. Το γεγονό ότι αυτέ οι πολύ μεγάλε τουριστικέ πόλει έχουν κάποια κινήματα απόρριψη του τουρισμού γιατί παρακολύουν την καθημερινότητα και ε, δημιουργούν ε, προβλήματα στι μεγάλε αυτέ πόλει. Και επίση ο τουρισμό κρουαζιέρα. Ο τουρισμό κρουαζιέρα σίγουρα αποτελεί μεγάλο εμ σημείο ε, τουρισμού και εσόδων για τη χώρα στην οποία σταματούν τα κρουαζιερόπλια, αλλά δημιουργούν ε, και επίσης ε, ε κάποια θέματα, ε, διότι θεωρείται ότι δεν ξοδεύει πολλά ο τουρίστας που φτάνει με το κρουαζιερόπλιο, γιατί είναι αυτάρκης λόγω του, του κρουαζιερόπλιου. Πρέπει να δούμε ε, όμως πώς μπορούμε να είναι επιτυχημένος αυτός ο τουρισμός, διότι αφορά και τις ανθρώπινες σχέσεις και πολλά άλλα πράγματα. Ευχαριστώ κύριε Ντεγκράντε και κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω για τη μελέτη η οποία πράγματι περιλαμβάνει πάρα πολλές πληροφορίες και εμένα μου ε, προξένησε το ενδιαφέρον μια πληροφορία που δεν περιλαμβάνεται και θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον ε, θα το εξετάσετε αυτό διότι είστε ε, Είμαι στην Επιτροπή Αλληλείας και στην Επιτροπή Μεταφορών. Το θέμα της ανάπτυξης του τουρισμού και του ναυτικού τουρισμού πρέπει να ε, συνδυάζεται και με κάτι το οποίο κάνει τουλάχιστον τμήμα της ομάδας μου και εγώ η ίδια, ε, τη διαφοροποίηση του τομέα της αλληλείας. Ένα τομέα ο οποίος τα τελευταία χρόνια βιώνει δυσκολίες για διάφορους λόγους, ε, μείωση των ποσοστώσεων, ε, έλλειψη ατόμων που θέλουν να ασχοληθούν με τον κλάδο αυτό κλπ. Πάρα πολλοί λοιπόν από τον ελληνικό τομέα μας ζήτησαν να τους βοηθήσουμε για τη διαφοροποίηση του κλάδου ώστε να μπορέσουν να ε, περιληφθούν σε αυτό το λεγόμενο ναυτικό τουρισμό. Και εμένα μου έκανε εντύπωση που δεν κάνατε ούτε μία αναφορά όταν αναφερθήκατε στις συνέπειες, στις θέσεις απασχόλησης, ε, τα προβλήματα και τις συστάσεις ε, στην ανάλυση αυτή και θα ήθελα να ξέρω αν υπάρχει κάτι τέτοιο, αν προβλέπετε να γίνει κάτι τέτοιο, διότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πώς ο ναυτικός τομέας συμβάλλει με θετικό ή με αρνητικό τρόπο ίσως στον αλληλευτικό τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μάιστερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη. Ε, ακούστηκε σαν θαραλέα, όχι σύντομη θα είμαι. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω για την παρουσίαση. Θα ήθελα να μας τη δώσετε, ίσως θα μπορούσατε να τη στείλετε σε όλους. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Και δεύτερον, ο ναυτικό τουρισμό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι τμήμα και του θεματολογίου της γαλάζια ανάπτυξη. Εγώ είμαι υπέρ τη ολοκληρωμένη θαλάσσιας πολιτική και συμβάλλει αυτό και στη γαλάζια ανάπτυξη. Ε, υπάρχουν μεγάλα ωφέλη από τον ναυτικό τουρισμό και στον κόσμο αρέσουν τα σκάφη. Αλλά φυσικά υπάρχουν και προκλήσει ε, και για περιβαλλοντικά θέματα, ε, για χωροταξικό σχεδιασμό ε, σε επίπεδο θαλάσσης κλπ. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά και ενδιαφέρει και την Επιτροπή Μεταφορών και καλό είναι να έχει άποψη η Επιτροπή Μεταφορών για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Τσέλισκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ίσως οφείλεται και στην άγνοιά μου και το γεγονός ότι είμαι και από μια χώρα χωρίς ε, θάλασσα. αλλά η μελέτη και οι παρατηρήσεις μου φάνηκαν ε, πολύ ενδιαφέρουσες για μένα. Δηλαδή αυτό είναι απλώς ένας ακόμα τρόπος μεταφορών και δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να θεωρείται κάτι διαφορετικό από τα αυτοκίνητα ή τα αεροπλάνα. Εδώ δεν αναφέρομαι μόνο στον ε, τουρισμό αλλά και την ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων και υπηρεσιών. Και πραγματικά μου φαίνεται λίγο παράλογο να είναι κάποιος για παράδειγμα κυβερνήτης σε σκάφος από την Κροατία και να παρέχει υπηρεσίες ε, και στα ύδατα της Ιταλίας ή στις ακτές της Ιταλίας αλλά δεν μπορεί κάποιος να αναβλώσει το ίδιο σκάφος ε, στην Ιταλία αλλά πρέπει να αναβλωθεί στην Κροατία. Τέλος πάντων είναι παράδειγμα, δεν αφορά τις χώρες, αλλά μου δημιουργεί έκπληξη. Δεν είναι θέμα του σκάφους ε, και των δεξιοτήτων σου, αλλά και των υπηρεσιών που παρέχεις. Ε, οι συνέπειες για τον τουρισμό ε, είναι πολύ σημαντικές. Κάθε άλλο παραμελητίες είναι τουρισμός ο οποίος αφορά και πολλά άτομα. Δεν μπορεί κάποιος να αναβλώσει για παράδειγμα ένα γιότ το 20 ατόμων. Χρειάζεται και προσωπικό στο σκάφος, επομένως είναι και ακριβώς τουρισμός αυτός. Βλέπω όμως μια έλλειψη φιλοδοξίας. Δεν ξέρουμε τι να κάνετε. Ορισμένες φορές ε, αναφερθήκατε στο αν υπάρχει ανάγκη. Εγώ θα ήθελα να σας καλέσω να είστε λίγο πιο φιλόδοξοι, να έχετε κάποιο πολιτικό στένος και να κάνετε κάποιες προτάσεις που να άρουν τους φραγμούς αυτούς. Θα βρείτε υποστήριξη στο Κοινοβούλιο με όλες τις ε, συνέπειες βέβαια, τις οποίες θα εξετάσουμε. Δεν θα ήθελα εδώ να θεωρήσω ότι είναι αμεληταία αυτά τα πράγματα. Η κυρία Αρνατού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κατάλαβα από το έγγραφο εργασίας ότι θέλετε να ενοποιήσετε τις άδειες ε, των επαγγελματιών ε, ε, Θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να είναι κρατικό και τελικά εσείς θέλετε να αυξήσετε το κοινωνικό ντάμπινγκ και σε αυτό το τομέα. Πάρα πολλοί ιδιοκτήτες ε, σκαφών ε, προτιμούν να έχουν σημαίες σε φορολογικούς παραδείσους και τώρα εσείς θέλετε να εργάζονται παντού χωρίς δυσκολία και σκύπερ από χώρες ε, ε, οι οποίοι δεν έχουν πάρει τις ίδιες άδειες, παίρνουν άδειες σαν κάποιους ανθρώπους που οδηγούν σκάφη στην, σε κάποιες χώρες. Το ίδιο κάνετε και με τους επαγγελματίες οδηγούς για παράδειγμα, με τους Πολωνούς οδηγούς Νταλίκας. Θα δημιουργήσετε δηλαδή τα ίδιες συνθήκες και στον τομέα των σκαφών. Υπάρχει και το θέμα της επικουρικότητας στον τομέα της ναυτιλίας. Εδώ πρέπει να το λάβουμε υπόψη, διότι ε, κάθε χώρα έχει τελείως διαφορετικές ανάγκες και λόγω κλιματικών και ωκεανογραφικών συνθήκων ε, και είναι ορισμένες φορές ε, ριζικά διαφορετικές αυτές οι ανάγκες. Πρέπει είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες του κάθε τομέα και να υπάρχει συγκεκριμένη εμπειρία στον τομέα. Ευχαριστώ πολύ. για ένα λεπτό να δώσω το λόγο στον εισηγητή. Ο κύριος Λάιναμαν έχει το λόγο για να κλείσει τη συζήτηση. Ναι, ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Η κυρία Μπιλμπάο ανέφερε ε, κάποια θέματα. Δεν θα μιλήσω για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την πολιτική της για το σεξ και το αλκοόλ. Θα περάσω στα επόμενα ζητήματα. Η ρύθμιση της αλίας και η αλία γενικότερα αναφέρεται σύντομα στο έγγραφο εργασίας, στο υπηρεσιακό αυτό έγγραφο και πραγματικά εκτιμούμε την μελέτη που έκανε η Επιτροπή Αλίας για το ρόλο του τομέα και τον αναδυόμενο ρόλο που έχει να παίξει. Επίσης, σε αυτό το υπηρεσιακό έγγραφο αναφέρεται ότι στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας υπάρχει ένα συγκεκριμένος φάκελος για το CLLD που είναι για την τοπική ανάπτυξη των κοινωνιών. Είναι ακριβώς αυτό που αναφέρατε. Μία διαφοροποίηση στο επάγγελμα των αλλιέων. Ε, περιλαμβάνει και τουριστικές δραστηριότητες γαστρονομικές περιηγήσεις ε, σε διάφορα εστιατόρια, αφού έχεις κάνει μια βόλτα με ένα σκάφος σε πολλές παράκτης περιοχές της Ευρώπης. Αν θέλετε μπορούμε να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα. Κυρία Μάιστεν, σε ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια σχετικά με την ατζέντα. Το εκτιμώ. Κύριε Ντελίτσια, είπατε προηγουμένως ότι Ε, ε, ακούσατε μάλλον από τον συνάδελφό σας ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα που θα πρέπει να τεθούν εάν ποτέ καταθέσει η Κομισιόν κάποια τέτοια πρόταση και γι' αυτό η μελέτη εξετάζει πολλέ επιλογές. Η νομοθεσία σε αυτό τον τομέα θα ήταν ιδιαίτερα περίπλοκη υπόθεση. Εν τούτης, εργαζόμαστε επί της εναρμόνισης των αδειών, για παράδειγμα, για να υπάρχουν κάποια κοινά στάνταρτ και μετά πέρα από αυτά να μπορούμε να προσθέτουμε κάποιου προσόντα, δηλαδή κάποιες απαιτήσει για συγκεκριμένα ε, θαλάσσιες συνθήκες, ε, γνώση του τοπικού περιβάλλοντος, των ντόπιων θαλασσών κτλ. Μιλήσαμε γιατί μιλήσατε για το πώς ε, εμποδίζουμε την εσωτερική αγορά. Ε, το είπα σύντομα, αλλά αναφέρεται στο εγγραφό μου πώς συμβαίνει, μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Πάμε στο επόμενο θέμα. Αυτό κλείνει. Έχουμε την έκθεση σύσταση για την ε, συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών για τις αεροπορικές υπηρεσίες. Εκθέση Γκρίφιν. Ε, νομίζω ο κύριος Βίλσον θα εκπροσωπήσει την κυρία Γκρίφιν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Εγώ εκπροσωπώ την κυρία Γκρίφιν, η οποία δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ, γιατί έχει μια συνάντηση σκιονδών εισηγητών. Από το 2003 υπάρχει συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών που αφορά τις εναέριες μεταφορές και αυτή η συμφωνία είναι μια πολύ τυπική συμφωνία η οποία αφορά κυρίως τομείς και θέματα που απορρέουν από την συνθήκη της Λισαβόνας. Μπορείτε στο κείμενο να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Η θέση της κυρίας Γκρίφιν είναι η εξής, ότι πρέπει να στηρίξουμε την συμφωνία αυτή. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Νίλσον. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο, η κυρία Βαντεκάπ. Ο κύριος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ευχαριστώ. Συμφωνώ απολύτως ε, με την εισηγήτρια και με τον ε, κύριο Νίλσεν. Μπορούμε να στηρίξουμε και να γνωμοδοτήσουμε θετικά Ήδη το 2000, όταν δεν υπήρχε τέτοιο κείμενο, η ενέργεια κυκλοφορία μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτών ήταν το 61% της συνολικής ενέργειας κυκλοφορίας. Σήμερα έχουμε πάει στο 35%. Έχουμε μια θεαματική πτώση. Γιατί, διότι βλέπετε ότι με τις διμερείς συμφωνίες με τις εταιρείες του κόλπου, παραδείγματος χάρη, έχει μετατοπιστεί ένας μεγάλος αριθμός των στόλων σε άλλες περιοχές. Την ίδια ώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν σημαντική προσπάθεια από μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών έτσι ώστε να ε, άρουν κάποιους περιορισμούς. Γιατί μετά την δημόσια διαβούλευση που οργανώνει το Κογκρέσο στις Ηνωμένες Πολιτείες τα πράγματα φαίνεται ότι θα αλλάξουν. Εμείς στην Ευρώπη δεν θέλουμε να αλλάξουμε απολύτως τίποτα. Και παραδείγματο χάρη, τι θα γίνει με αυτή την απαγόρευση λάπτοπ. Θα συνεχίσουμε με αυτό ή θα το αλλάξουμε. Κυρία Φώστερ, όχι. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι στις 21 Νοεμβρίου στις 2. Η Επιτροπή. Όχι. Allez, on continue. Et on va demander... Το επόμενο θέμα είναι και κλεισμένων των θυρών. Σας παρακαλώ πολύ, όποιος ε, δεν ανήκει στην Επιτροπή να εγκαταλείψει την αίθουσα.